Okay, Λοιπόν, κύριε και κύριοι, ζητώ συγγνώμη, αλλά μου το είπε και ο Αντώνιο ότι εδώ πέρα τα σανσέρ στα κτίρια του Κοινοβουλίου είναι και το χάος. Ε, ε, λέψαμε, είδαμε και πάθαμε για να φτάσουμε. Ζητώ συγγνώμη και πάλι και περνούμε στην απογευματινή συνεδρίαση. Θα δώσουμε το λόγο και στον κύριο Επίτροπο και στον κύριο Ρούτε, αλλά πρώτα στον Επίτροπο. Είναι σε αυτού αφιερωμένο το απόγευμα για την παρουσίαση της δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και μετά την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε Σίμψον, είναι χαρά μου να σας παρουσιάσω το λεγόμενο τέταρτο πακέτο των σιδηροδρόμων που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν στα τέλη του Ιανουαρίου. Είναι σημαντικό και φιλόδοξο το πακέτο αυτό. Ε, αποτελείται από μια γενική επισκόπηση μια γενική ανακοίνωση πάνω στην νομοθετική πρόταση, τρει ε, μελέτες αδικτύπου, τρει εκθέσεις και τρία έγγραφα εργασίας του προσωπικού. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Σιδηροδρόμων για να παράσχουμε καλύτερη ε, ποιότητα στις ε, σιδηρομικέ υπηρεσίες. Προτού να μπω σε λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να πιω ένα καφέ. Να σας πω ε, κάποια γενικά πράγματα που είπα στην ε, ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε όλους μας αρέσουν οι σιδηρόδρομοι και στον Bismarck αρέσανε και στη σύγχρονη εποχή μας αρέσουν, αλλά οι σιδηρόδρομοι περνάνε παρακμή. Είχαμε πτώση στη μεταφορά ε, αγαθών ε, από 11,5% ε, το 2000 σε 10,2% σήμερα. Είδαμε σημαντική μείωση στη χρήση από το 1990. Οι σιδηρόδρομοι απαιτούν και περισσότερα χρήματα των φορολογούμενων 46 δισεκατομμύρια το 2009 και δεν είναι όλες οι χώρες ε, σε θέση ε, να κάνουν τις επενδύσεις αυτές. Επίσης, ε, στη Γαλλία οι σιδηρόδρομοι έχουν συσσωρεύσει 28 δισεκατομμύρια χρέους, το ίδιο στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο. Ε, και 900 παραγωγούς, κατασκευαστές ε, εξοπλισμού έχουμε, ε, αλλά λόγω της παρακμής των ευρωπαϊκών συνδρόμων δεν μπορούν να πουλήσουν στην Ευρώπη τα προϊόντα τους. Οι επενδύσεις αυξάνονται στην Ασία, το Μέση Ανατολή, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται λοιπόν και για εξαγωγική αγορά. Σήμερα στις ειδήσει είδα ότι η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία ανακοίνωσαν ότι θα κατασκευάσουν ε, ε, ανάμεσα στην ε, Σιγκαπούρη και την Κουάλα Λουμπούρ συνδρομική γραμμή ψηλής ταχύτητας. Αλλά οι εξαγωγές είναι δύσκολες εάν δεν λειτουργεί καλά και η εσωτερική αγορά σημαντικό ερώτημα, το οποίο μάλλον έχετε συζητήσει και εσείς ε, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της Λευκής Βίβλου. Ε, το ερώτημα λοιπόν είναι, ε, όταν συζητάμε το πακετό σιδηρόδρομων, χρειαζόμαστε τους σιδηροδρόμους, διότι ε, υπάρχει και η άλλη άποψη. Η άλλη άποψη είναι να αναπτύξουμε τις ε, οδικές ε, μεταφορές. Ε, οι αυτοκινητοβιομήχανοι αυτή τη θέση υποστηρίζουν. Και αντί για διευρωπαϊκά δίκτυα και τις προτεραιότητες ΕΣΕΦ να χτίσουμε αυτοκινητόδρομους στην Ανατολική Ευρώπη και να έχουμε διασυνοριακούς, διασυνοριακές οδικές αρτηρίες. Ε, αλλά ε, η άποψη αυτή δεν απαντάει στο πρόβλημα της ε, συμφόρησης που αφαιρεί ένα εκατομμύριο σε αέπανα χρόνο και χάνουμε και πολλές ε, ζωές ε, το χρόνο στις οδικές μεταφορές, ενώ από τους δρόμους χάσαμε μόνο 62 το 2012. Και βέβαια δεν μπορούμε ούτε να ε, ονειρευόμαστε τους στόχους μας περί ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής εάν βασιστούμε στις οδικές μεταφορές. Πολύ σημαντικό λοιπόν στο πακέτο αυτό είναι ότι εάν δεν έχουμε μια σωστή πολιτική μεταφορών για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, οι σιδηρόδρομοι θα είναι απλά παιχνίδι πολυτελείας για τους πολίτες των πλουσίων χωρών. Δεν θα έχουμε πανευρωπαϊκό σύστημα, δεν θα έχουμε ε, ενιαία αγορά, δεν θα έχουμε ε, μια, ε, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο σιδηροδρόμων. Το πακέτο που προτείνουμε σήμερα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτα να εξαλείψουμε τους ε, διοικητικούς ε, και ε, και τα γραφειοκρατικά εμπόδια με τη διαλειτουργικότητα. Να ανοίξουμε τι εσωτερικές, τις εγχώριες αγορές, να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση της διαχείρισης υποδομών. Υπάρχουν ελλείψεις στο παρόν σύστημα όσον αφορά την πιστοποίηση των οχημάτων. Ε, σχεδόν 11.000 ε, ε, κανόνες υπάρχουν, εμπορική τεχνική και ασφαλεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πιστοποίηση και τη διάθεση στην αγορά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες για όλους τους οικονομικούς φορεί και να διασφαλίσουμε ίσα δικαιώματα πρόσβασης το αποκεντρωμένο σύστημα ε, εθνικών αρχών ασφαλείας ε, δημιουργεί ε, κάνει πολύπλοκη την πρόσβαση στην αγορά για παράδειγμα, ε, μηχανές ε, σιδηροδρόμων ε, εγκεκριμένες στη Γαλλία και στην Βρετανία δεν μπόρεσαν να εγκριθούν σε άλλη χώρα λόγω της θέσης, της, λόγω της, της θέσης, το που βρισκόταν η θέση του οδηγού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας ε, ώστε να μπορεί κανείς ε, να λειτουργήσει όλη την Ευρώπη. Θέλουμε κανόνες ε, διαλειτουργικότητας ώστε να έχουμε εξοικονόμηση κλίμακας να μειώσουμε το, κόστος, το διοικητικό κόστος και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να αποφύγουμε τις διακρίσεις. Αυτός είναι ο λόγος για την πρόταση της ε, Επιτροπής ε, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες πιστοποίησης ε, και για τις επιχειρήσεις και για τα οχήματα. Έτσι θα διασφαλίσουμε την διασυνοριακή λειτουργία. Θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά με δύο τρόπους. Πρώτον, με δικαίωμα πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες προς τους ε, και με ε, τον ανταγωνισμό εντό τη αγορά. Η μελέτη αντικτύπου τη Κομισιόν δείχνει ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, θα έχουμε καλύτερη αποτελεσματικά των υπηρεσιών και το τα πλεονεκτήματα ε, εάν ανοίξουν οι, οι αγορές υπολογίζονται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2035. Η Κομισιόν πρότεινε να ανοίξει τις εγχώριες ε, αγορές ε, σιδηροδρόμων στον ανταγωνισμό, αλλά βαθμιαία. Επίσης, τα προνόμια των κρατών μελών και των αρχών τους να καθορίζουν τις ε, υποχρεώσεις ε, στην ε, εσωτερική αγορά, στην χώρια αγορά θα διατηρηθεί. Θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων πρόσβαση σε όλες τις υποδομές της Ευρώπης χωρίς διακρίσεις. Το άνοιγμα τη αγορά θα πραγματοποιηθεί βαθμιαία και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτές ε, διαδικασίες ε, διεξαγωγή διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, η δυνατότητα απευθεία ανάθεσης που υπάρχει σήμερα δεν θα τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, σε περίπτωση συμβάσεων μικρής κλίμακας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε επίγουσες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών. Επίσης η πρότασή μας ε, θέλει να ωφελήσει τους ε, επιβάτες, ενθαρρύνει ε, λοιπόν τα κράτη-μέλη και τις σχετικές επιχειρήσεις να σκεφτούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων με τρόπο μη διακριτικό για όλες, για όλες τις επιχειρήσεις ιδεοδρόμων. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα στοιχείο που έχει να κάνει με το άνοιγμα των εγχωρίων αγορών, την κοινωνική πτυχή. Εάν βελτιώσουμε την, ε, εμπιστοσύνη, την, ε, συγγνώμη, την ελκυστικότητα των σιδηροδρόμων, θα έχουμε περισσότερους ε, επιβάτες, το οποίο σημαίνει θα θα χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή η έλλειψη προσωπικού είναι, κάτι που μας απειλεί και έχουμε δει σε άλλες χώρες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Εάν αλλάξει μια σύμβαση και μεταφερθεί από έναν ε, πάροχο σε έναν άλλον, ε, τότε οι δημόσιες ε, αρχές, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διασφαλίσουν την μεταβίβαση και του προσωπικού και τη διασφάλιση κοινωνικών προτύπων. Η Κομισιόν θέλει να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση της υποδομής ε, διασφαλίζοντας ε, μια σειρά λειτουργιών που βελτιστοποιεί την ε, χρήση της υποδομής. Όλες οι σχετικές λειτουργίες αναφέρονται στην πρόταση. Βλέπετε τη διαφάνεια που δείχνει την δομή διακυβέρνησης στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πιο δύσκολο θέμα είναι οι κάθετες δομές ε, και σημείο κίνησής μας ε, είναι ότι η πιο αποτελεσματική λύση για να διασφαλίσουμε το δίκαιο ανταγωνισμό και την μη διακριτική μεταχείριση είναι ο διαχωρισμός ε, των θεσμών. Αυτό πρότεινε η Κομισιόν στον τομέα της ενέργειας και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και εδώ. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανείς νέες δομές όταν θα έχει τεθεί σε ισχύ η πρόταση. Θέλουμε δηλαδή ε, σε περίπτωση ε, δεν θα μπορούν να δημιουργηθούν νέες ε, εκμεταλλεύσεις χαρτοφυλακίου, holding structures και θα υπάρχουν χέγγια ώστε να έχουμε ίσες ε, συνθήκες για όλους ε, τους ε, οικονομικούς φορείς. Τα εχέγγυα αυτά βασίζονται στην απέτηση περί διαχωρισμού που ήδη ισχύουν από το 2003 σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πείρα μας δείχνει ότι οι υποχρεώσεις αυτές είναι πολύ γενικές και δεν εφαρμόζονται σωστά. Ε, έτσι βλέπουμε ακόμα διακριτική μεταχείριση εντός του τομέα των και η πρόταση της Κομισιόν προτείνει να διασαφινιστούν τα ε, συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ε, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των υποδομών. Τα εχέγγυα αυτά ε, αντικατοπτρίζουν μια συμβαστική πρόταση που είδαμε στον τομέα των σιδηρόμων πριν τρία χρόνια. Προσπαθήσαμε όμως να απλοποιήσουμε τους κανόνες ώστε να αποφύγουμε ε, την περίτη γραφειοκρατία. Θα ήθελα να αναφέρω και άλλες ε, σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη διακυβέρνηση των υποδομών. Όλοι οι οικονομικοί φορείς καθώς και οι νέοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν με για την ε, ε, διαχείριση των υποδομών. Επίσης, προτείνουμε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο ε, διαχειριστών υποδομής, ώστε να έχουμε ευρωπαϊκή υποδομή. Είμαι βέβαιος ότι η πρόταση της Κομισιόν βρίσκει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία που χρειάζονται κάποια κράτη-μέλη για να διατηρήσουμε να διατηρήσουν τις παρούσες εκμεταλλεύσεις τους και να έχουμε Πιστεύω επίση ότι έχουμε τα απαραίτητα χέρια για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία, ε, το, το, διαχωρισμό των υποδομών, το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσουν σωστά οι σιδηρόδρομοι. Όπω σα είπα, είναι ε, φιλόδοξο το πακέτο αυτό. Περιμένει ο σιδηροδρομικό τομέα εδώ και πολλά χρόνια, ε, όπω και οι οικονομικοί φορεί και πιστεύω και οι ε, επιβάτε, το πακέτο αυτό εδώ και πολύ καιρό. Η Κομισιόν θέλει να ε, συνεργαστεί επικοδομητικά με του νομοθέτε ε, για να ε, ε, υιοθετήσουμε το πακέτο αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ευαίσθητα θέματα, υπάρχουν τοπικές ανησυχίες. Η Κομισιόν βασίζεται ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να διασφαλίσει να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα σύνδρομων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Επίτροπε αρχίσω από τους συντονιστές Γκρός, Ελχαντράου, Ιντεμπάκερ, από τους φιλευτέρους και κύριος Κράμερ. Και μετά Ρικέ, Λάιχτφριντ, Σαβισάρ, Πίρκερ, Μπαχ, Καντσάν, άλλος κανείς, Φλέκενστάιν. Mr. Tremosa. Okay. Hey. Okay, Καλώς. Αρχίζουμε λοιπόν. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση του πακέτου αυτού, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε από διάφορες οδούς και να πληροφορηθούμε. Χαιρόμαστε όμως που μας το παρουσιάζει και επίσημα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τούτο εδώ το Κοινοβούλιο αγωνίζονται εδώ και χρόνια για να έχουμε αποτελεσματικούς, αποδοτικούς σιδηροδρόμους στην Ευρώπη. Αυτή είναι και η στόχη μας και πιστεύουμε ότι στις εμπορευματικές μεταφορές και στις μεταφορές γενικότερα ε, ο σιδηρόδρομος μπορεί να παίξει ένα ρόλο πιο πρωταγωνιστικό από αυτό που κατέχει αυτή τη στιγμή. Ρωτώ, είναι και το Συμβούλιο πεπισμένο γι' αυτό? Γιατί βλέπω τις τελευταίες αποφάσεις για τα οικονομικά και ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών ήταν καλό το πρόγραμμα και το σχέδιο με ιδιαίτερη μέρημνα για το σιδηρόδρομο και πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Συμβούλιο ε, δεν ε, ακολουθεί απολύτως τον ίδιο δρόμο. Επίσης γνωρίζουμε και στο παρελθόν ότι χωλαίνει η εφαρμογή. Ε, χρειάζεται και μια δεκαετία και παραπάνω για να εφαρμοστούν με επιτυχία. Και επειδή συζητήσαμε και αποφασίσαμε μια αρχή ε, ελεκτική και ρυθμιστική που πρέπει να είναι ανεξάρτητη και για μένα ήταν εκ των όνου κάνευ για να είναι πιο αποτελεσματικά τα όσα προτείνονται σε αυτή τη δέσμη ή σε κάποια άλλη αναπροσαρμοσμένη. Θα ήθελα να τα πω λοιπόν αυτά εισαγωγικά και να στείλουμε και ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο. Έρχομαι τώρα στην πρόταση και το σύνολο πακέτο και τη δέσμη των μέτρων αυτών. Αλλά σήμερα δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες και ιδιαίτερα εξ ονόματος της ομάδας μου, να τονίσω μόνο τρία πράγματα. Πρώτον, χαιρόμαστε πάρα πολύ και καλωσορίζουμε την πρόταση για την τεχνική διαλειτουργικότητα και συμβατότητα των δικτύων. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι παραλογισμοί στις συμπεριφορές που παραμένουν σήμερα. Υπάρχουν σύνορα ακόμα πραγματικά στο σιδηρόδρομο και πρέπει αυτά να σταματήσουν. Γι' αυτό διαλειτουργικότητα, συμβατότητα και ενισχυμένος οργανισμός για να είναι ανταγωνιστικός και αυτός ο τρόπος και αυτό το μέσο μεταφοράς για να μπορούμε να ε, λειτουργούμε καλύτερα σε σχέση με τα όσα σήμερα υφίσταται σιδηρόδρομος. Μετά, τι περιμένουν οι πολίτες. Έχουν προσδοκίες για την παροχή υπηρεσιών. Και αν δούμε το σιδηρόδρομο, ε, είναι ο πιο μισητός, αγαπημένος ε, πολλών ανθρώπων. Γιατί πολλοί αγαπούν το σιδηρόδρομο, αλλά τον υπονομεύουν, τον ε, υποτιμούν κάθε φορά μπορεί ο σιδηρόδρομος να είναι και πιο ασφαλής και πιο καθαρός, αλλά ίσως δεν είναι αρκετά αξιόπιστο μέσο μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί περισσότερο και η ε, αξιοπιστία του ως μέσο μεταφοράς. Έρχομαστε σε ένα πολύπαθο θέμα, ε, παλιό, του διαχειριστή της ε, υποδομής, με, του δικτύου δηλαδή, με εκείνον που κάνει τα δρομολόγια. Αυτό είναι όπως τη λογοτεχνία, τα παλιά δράματα και τραγωδίες. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες. Ε, των κρατών μελών και ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Το φανάρι είναι άλλες φορές κόκκινο, άλλες φορές πράσινο, κίτρινο αλλά ε, θα πρέπει αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι η αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη λειτουργία και όχι ένα οποιοδήποτε δόγμα. Αν ξεφύγουμε από τα δόγματα και τις αγκυλώσεις αυτές θα ε, προχωρήσουμε. Και βεβαίω να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού αλλά και διαφάνεια να κυριαρχεί για να μην ε, καταργηθούν τελείως οι λεγόμενες εγκάρσεις ή πλάγιες επιδοτήσεις, ε, γιατί χρειάζονται βεβαίως καμιά φορά και κρατικές ενισχύσεις, αλλά και η λειτουργία ε, των επιχειρήσεων. Και επίσης ο σιδηρόδρομος μπορεί να διαφυλάξει, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και μάλιστα ποιοτικέ. Αυτά. Άκουσα και το είδα το σφυράκι που με απειλεί. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά ως ΕΛΚ θέτουμε προσυζήτηση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ ο κύριος Χαντράουι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την εισαγωγή του. Αυτή τη φορά δεν θα μιλήσω για τη διαλειτουργικότητα και την ενίσχυση του ρυθμιστή. Τα είπατε πολύ ωραία, ούτε για τις δομές, τα είπαν και θα τα πούνε και άλλοι συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε κάτι που έχει σημασία για την πλειονότητα των πολιτών μας και αυτό είναι η παροχή υπηρεσιών. Ο στόχος ποιος θα είναι, να έχουμε περισσότερους επιβάτες στο σιδηρόδρομο και να είναι καλές οι συνθήκες με μεγάλες ε, οι προσφορές και για μικρότερες διαδρομές και δρομολόγια όχι τόσο δημοφιλή, τόσο συχνά. Γιατί η ομάδα μου ανησυχεί και θέλω να σας ρωτήσω για δύο πράγματα. Ε, για την απελευθέρωση και για τις συμβάσεις ε, με το δημόσιο. Open access το λέτε αυτό, ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο. Ναι, και μετά όμως έχετε και συμβάσεις για τη δημόσια υπηρεσία κοινοφιλή ουσιαστικά η υπηρεσία είναι αυτή. Με δημόσια συμβάσει. Αν εγώ είμαι επιχείρηση όμως και θέλω να κάνω μια προσφορά για μια δημόσια σύμβαση, θα πρέπει να δω και τι ε, υπηρεσίες προσφέρω, αλλά και τι ανταμοιβή παίρνω για τις υπηρεσίες αυτές σε ένα ε, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τη σύμβαση. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια προβλεψιμότητα σε όλα αυτά. Εσείς όμως αυτό το καταργείτε περίπου, διότι ε, επιτρέπεται να ε, υπάρχει ανταγωνισμός από το ε, σύστημα Open Access ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη περιφέρεια ε, που θα έρθουν και θα διαλέξουν τις πιο κερδοφόρες γραμμές, ας πούμε, κάποιοι εξωτερικοί και θα κάνουν αυτά τα δρομολόγια καθένα θα διαλέγει το πιο κερδοφόρο ε, κομμάτι και αντίστοιχα θα είναι και η τιμολόγηση του εισιτηρίου. Έτσι δεν είναι. Ποιε είναι λοιπόν οι δυνατότητε εκεί και ο ρυθμιστή πώ θα τα ελέγχει και θα ρυθμίζει και θα ε, περιορίζει τον ανταγωνισμό. Πολύ ασαφή μα τα λέτε. Ένα άλλο θέμα. Οι συμβάσει αυτέ οι δημόσιε για παροχή υπηρεσιών κανονικά αυτό πρέπει να αφορά μικρές περιοχές, αστικές περιοχές ας πούμε. Και λέτε ε, το πολύ 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα σιδηροδρόμου ή ένα τρίτο της επικράτειας. Αλλά ο συνδυασμός διαφόρων ε, προϋποθέσεων που βάζετε εκεί και ορών μπορεί να σημάνει, σαν μια χώρα για το Βέλγιο, ότι θα πρέπει να σπάσουμε στα 8 το σιδηρόδρομο. Και μετά να αρχίσουμε να δούμε πώς θα βγει στην αγορά το κάθε 8 και πού είναι η παροχή υπηρεσιών και πώς βελτιώνεται η παροχή προς τον καταναλωτή και τον επιβάτη προκειμένου. Εγώ φοβούμαι ότι μάλλον θα προκληθούν περισσότερα προβλήματα παρά θα λυθούν και ζητώ μια λύση στα μέτρα του κάθε κράτους μέλους. Βεβαίως θέλουμε αποτελεσματικό σιδηρόδρομο αλλά και αποδοτικό, αλλά ο επιβάτης να υποφελείται και όχι να είναι σε χειρότερη μοίρα. Γιατί δεν είμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίως Ντεμπάκερ των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του και τη νέα πρόταση και το, τη ε, δέσμη. Είναι το τέταρτο πακέτο για το σιδηρόδρομο πλέον. Και εδώ στο Κοινοβούλιο είμαστε πεπισμένοι όλοι ότι μια ανοιχτή αγορά σιδηροδρόμων, ε, πιο αποδοτική από τη σημερινή ε, θα έχει ωφέλεια πολλαπλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε την πρόταση του Επιτρόπου και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία στην πρόταση αυτή για να μπορέσουμε και να τον ακολουθήσουμε ε, πλήρω Από πλευράς της ομάδας μου όμως θέλω να τονίσω και κάποια σημεία που δεν είναι ίσονος σημασίας. Να δούμε ποια είναι η ποιότητα των σιδηροδρόμων και πώς θα αυξηθεί για να προσελκύσει και περισσότερες ε, εταιρείες και περισσότερους επιβάτες και εταιρείε να το επιλέγουν ως εναλλακτική ε, μέθοδο μεταφορών. Ουσιαστικά τι είναι σιδηρόδρομοι σήμερα, είναι τα τελευταία κρατικά μονοπόλια που απομένουν ε, και δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός, ούτε αρκετή διάνοιξη, ούτε αρκετή διαφάνεια. Υπάρχει ένα πλαίσιο και μια δομή έχουν οι σιδηροδρομικές εταιρείε που χρειάζονται μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, θα πρέπει να ενισχυθεί ε, ο διαχειριστής ε, των υποδομών και να υπάρχει και ένα δίκτυο όλων αυτών των διαχειριστών των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω και την προσωπική μου γνώμη για το περίφημο unbundling την αποδέσμευση ε, χαιρόμαστε και ελπίζουμε η ε, πρόταση και ε, ο έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι αποτελεσματικός γιατί έχουμε διάφορα συνικά τείχη εδώ πέρα που κινδυνεύουν να υψωθούν. Θα πρέπει αυτά να τα αποφύγουμε. Έγινε λόγος για τις δημόσιες συμβάσεις, για την κοινοφιλή υπηρεσία. Βέβαια, θα πρέπει να είναι και ποιοτική υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό. Άκουσα το Ματιό Γκρό και συμφωνώ και εγώ ότι έχει μια σχέση αγάπης μίσους ο πολίτη με το σιδηρόδρομο. Ναι, αν υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια και με... Ε, αν ε, κοβόταν και λίγο το λίπος που υπάρχει στις σιδηροδρομικές εταιρείες, ε, θα υπήρχαν μεγαλύτερες δυνατότητες και για τις μεταφορές και καλύτερη εξυπηρέτηση και των επιβατών. Ε, σε ό,τι αφορά τη τιμολόγηση του εισιτηρίου και κάποια άλλα σχετικά ε, μπορούμε ε, να συζητήσουμε περισσότερο. Και χαίρομαι επίσης που ο Επίτροπος αναφέρθηκε και σε μια κοινωνική πλαισίωση. Έχουν δείξει και οι μελέτες ότι όταν ανοίγει μια, εταιρεία, μια αγορά, συγγνώμη, ανεβαίνουν οι προδιαγραφές, δεν πέφτει το επίπεδο παρά όσα πιστεύουν ορισμένοι. Η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς βοηθάει για διαφάνεια, για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και, εν πάση περιπτώσει, οι κοινωνικές ε, προδιαγραφές δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μειώνονται ε, και πέφτει το επίπεδό τους. Ε, καλές οι προτάσεις, θα συζητήσουμε τα διάφορα επιμέρους στοιχεία και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη με έναν Ευρωπαίο ρυθμιστή, γιατί στο παρελθόν υπολείποντο τις προσπάθειες αυτή και Καλό είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρόμων και είναι επίγουσα ανάγκη και για τους πολίτες και για τις εταιρείες μας. Ο κύριος Κράμερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Σιδηροδρόμων. Ε, όλοι το θέλουν εδώ, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη ε, βλέπουμε ότι έχουμε patchwork και με κενά στα σύνορα. Ε, από τις ε, εμπειρίες στην μεταφορά αγαθών. Είδαμε στις κάτω χώρες αύξηση 40%, στη Γερμανία 30%, ε, στην ε, Πολωνία 20% με το που άνοιξαν ε, τα σύνορα. Αλλά Εάν θέλουμε να δούμε τις ε, μεταφορές με, πολλά, με διάφορα μέσα, εκεί βλέπουμε τα μεγάλα ε, και να, εάν έχουμε ανταγωνισμό στο, στα σιδηρόδρομα ε, και δεν ασχοληθούμε με τους άλλους τομείς, τότε θα αποτύχουμε. Έχουμε τέλεια να χιλιόμετρα, έχουμε διόδια για τα για τα φορτηγά στους δρόμους, ε, ε, οι ε, αερομεταφορές για παράδειγμα δεν πληρώνουν φόρο για την κυροζήνη. Εάν δεν αλλάξουμε αυτές τις ανισότητες τότε θα αποτύχουμε γενικά και στα, ούτως ή άλλως χρήματα χρειάζονται και αυτό είναι αποφασιστική σημασία. Ε, κάναμε μια μελέτη και είδαμε ε, πού πηγαίνει το ευρωπαϊκό χρήμα. 60% στους δρόμους, 20% ε, στους σιδηροδρόμους. Δεν άκουσα τίποτα από εσά ε, σχετικά με αλλαγή της σηματοδότησης αυτής. Τουλάχιστον 40% στους σιδηροδρόμους, το πολύ 20% στις οδικές μεταφορές. Η χρηματοδότηση παίζει ρόλο στην, ε, φυσικά, διότι ε, στην τελευταία δημοσιονομική περίοδο θέλαμε 20 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Συμβούλιο τα μείωσε αυτό σε 8 δισεκατομμύρια, αλλά χωρίς να διαγράψει κανένα πρόγραμμα και το Connecting Europe ε, θέλουμε να ε, ε, υποστεί περικοπές, δεν τίθενται προτεραιότητες. Ο Μόντι και ο Λάντ συναντώνται και λένε ότι είναι σημαντική η γραμμή για το Τουρίνο ωραία, αλλά τελικά καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολλά προγράμματα ε, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αλλά δεν έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να το κάνουμε. Και θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε και τις ε, ε, χρηματοδοτικές ε, επιρροές. Επίσης αναφερθήκατε στην γραμμή του Κάρδη Ούλμ, 3 ε, δισεκατομμύρια στοιχείς, γι' αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά και με τα χρήματα αυτά ε, δεν ε, μπορείτε όχι να χρηματοδοτήσετε τη γραμμή από το Βερολίνο προς την Πολωνία, τρεις γραμμές. Ε, αυτό να κάνετε. Και τέλος, στην Γερμανία, επειδή οι επιχειρήσεις αποφασίζουν όλα, πάνω από 50% των χρημάτων που δίνουν τα κριτήρια για τις περιφερειακές για τις ε, ε, ε, περιφερειακές μεταφορές, όλα αυτά πάνε τελικά στους σε λάθος μέρη, το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ακριβές οι μεταφορές. Γιατί στοιχίζει στη Φραγκφούρτη 3 ευρώ η μεταφορά για το αεροδρόμιο και στο Βερολίνο 25 ευρώ. Εάν αυτό δεν είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ των οδικών μεταφορών, τότε εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα πρέπει να τα αλλάξετε όλα αυτά και ε, θέλουμε βέβαια αποτελεσματικότητα, χρειαζόμαστε όμως ε, και αποτελεσματικότητα στις ε, υποδομές. Η Κομισιόν τα περασμένα χρόνια, αλλά και εσείς εδώ σήμερα, αν δεν τα, αν να το κάνετε και αν δεν το κάνετε αυτό, τότε θα αποτύχουμε. Θα πρέπει να σκεφτείτε ολιστικά όχι μόνο τον συνδρομικό τομέα. Ευχαριστώ. Να ζητήσουμε από τον Επίτροπο να απαντήσει, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχω ακόμα 12 ώρες. Μπορώ να κάνω διαίρεση ακόμα. Εάν θέλετε λοιπόν να απαντήσετε στις πρώτες παρεμβάσεις, Επίτροπε, και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπου βουλευτές. Ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές και τους συντονιστέ. Φίξατε τα πλέον σημαντικά ζητήματα και θα προσπαθήσω να τα συγκεφαλαιώσω σε ομάδες σε σύνολα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα τεράστιο πακέτο, μια τεράστια δέσμη μέτρων, από τα μεγάλα. Και ξεκινήσαμε από το Ρίκαστ για τους σιδηροδρόμους, όταν σχεδιάσαμε το πακέτο, για να δούμε τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει. Και το πακέτο αυτό είναι περίπου όπως το είχαμε φανταστεί όλοι στις ομάδες σας είχατε την δυνατότητα να συναντηθείτε με τους εμπειρογνώμονές μας από τη Γενική Διεύθυνση MOVE για να δείτε τις λεπτομέρειες της αναδιατύπωσης. Διότι υπήρξαν πολλές λεπτομέρειες. Είχαμε λεπτομερείς ε, αναλύσεις και δεν είναι η τελευταία συζήτηση σημερινή από αυτές που θα γίνουν. Τώρα με το Συμβούλιο τι θα γίνει, το θίξατε και αυτό. Ε, το Συμβούλιο Περιλανδικής Προεδρίας θα συζητήσει στις 11 Μαρτίου πολύ σύντομα, γιατί ήταν ε, σημαντικό το πακέτο αυτό να εγκριθεί τουλάχιστον πριν το τέλος Ιανουαρίου, ώστε να δει τις προτάσεις και το Συμβούλιο. Θα δούμε τι στάση θα τηρήσουν, όμως είναι κάτι που το αναμένουμε. Ε, το πακέτο το ενημένουμε και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρξει επικοδομητική προσέγγιση. Δεν φανταζόμαστε πάντως να υπάρξει τεράστια αντίρρηση και αντίσταση για την όλη δέσμη, απλώς διαφορετικές τάσεις και τοποθετήσεις. Πολύ θίξατε το θέμα του Ιδρύματος για τους Ευρωπαϊκούς Σιδηροδρόμους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά αυστηρή σχετικά. Θέλουμε να ενδυναμωθεί ο οργανισμός των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, είναι κάτι το αναγκαίο τόσο ή άλλως και καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να πρικοδοτηθεί και με τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα. Νομίζω θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι απλή και ίσως με κάποιους δασμούς στην ε, όλη επιμηχανία. Το κεντρικό σύστημα αδειοδότησης ίσως είναι μία λύση. Τα τέλη πάντως θα μας βοηθήσουν. Με τους νέους σιδηροδρόμους, τις νέες αμαξοστοιχίες, η εξοδότηση θα κοστίζει 6 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια η επανέγκριση. Καταλαβαίνετε ότι ένα κεντρικό σύστημα θα μας ε, ωφελήσει ιδιαίτερα, θα ωφελήσει και τη βιομηχανία των σιδηροδρόμων, διότι είναι μεγάλο το τίμημα που καταβάλουν στο δομό των οικονομικών με όλη αυτή την πολύπλοκη δομή. Για τις υποχρεώσεις των κρατικών υπηρεσιών και την άνοιγμα, την απελευθέρωση των αγορών με τις τοπικές περιφερειακές αγορές και τους επιβάτες. Είμαστε ιδιαίτερα διαλλακτικοί στις προτάσεις αυτές. Πολλές από τις ε, ιδέες μας είναι και αρκετά μετριοπαθείς. Οπότε μπορούμε μπορούμε να συνδυάσουμε και να συμβιβάσουμε μεταξύ τους τις διαφορετικές εθνικές απόψεις. Ελπίζουμε ότι σταδιακά θα μπορέσουμε να οργανώσουμε το άνοιγμα της αγοράς, ώστε να μην γίνει κάτι το επαναστατικό και ξαφνικό. Όλα αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αλλά εμεί μπορούμε να φανούμε ευέλικτοι και διαλεκτικοί. Θέλουμε απλώ ένα σύστημα σφαιρική προσέγγιση, συνολικό που να λειτουργεί εύρυθμα. Τέθηκε και ένα μείζον ζήτημα από του περισσότερου από εσά ε, για του διαχειριστέ των υποδομών και τους ε, φορείς λειτουργίας. Η Επιτροπή προτείνει τον πλήρη διαχωρισμό, την ε, σαφή διάκριση μεταξύ των δύο. Εγώ να προσθέσω εδώ μία λεπτομέρεια. Στο πακέτο αυτό θέλουμε να υπάρχει μια σαφής προστιθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τι θα προκύψει αν έτσι διακρίνουμε τις υποδομές από τους φορείς που τις λειτουργούν. Θέλουμε να έχουμε σιδηροδρομικά δίκτυα. Να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί πανευρωπαϊκό, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Δεν μπορεί να έχουμε υποδομές, ε, βαγόνια και αμάξια τα οποία να καταβάλουν τέλη τα οποία να καταλήγουν στις τσέπες των ανταγωνιστών. Αυτό είναι τόσο απλά η συλλογιστική μας. Θα υπάρξουν τρόποι και μέθοδοι να καταπολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι αυτό ακριβώ. Και είναι ένα σημείο όπου δεν μπορούμε να φανταστούμε να υπάρξει συμβιβασμό. Δεν ήταν ε, το θέμα και δεν δυσκολευτήκαμε να δεχτούμε τους οριζόντιο, την οριζόντια διοργάνωση, αλλά είναι, πρέπει να είναι σαφή οι κανόνε διαχωρισμού μεταξύ των διαχειριστών των υποδομών και όσων λειτουργούν τι υποδομέ. Πρέπει να είναι οι ροέ των κονδυλίων σαφείς, διαφανείς και να μπορούμε να τι παρακολουθήσουμε. Αυτό πρέπει να το ε, συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στάση από την οποία θα ξεκινήσουμε. Οπότε ναι, Μπορούμε να δεχτούμε και την οριζόντια διοργάνωση, αλλά είναι άλλο πράγμα η διάκριση των διαχειριστών των υποδομών και όσους ε, είναι οι φορείς που λειτουργούν τις υποδομές, αλλά αυτό θα πρέπει επίσης να έχει να κάνει με την διαφανή διαχείριση των ροών χρημάτων. Δεν μπορεί κάποιο που είναι ιδιοκτήτη των υποδομών να είναι ο ίδιο και φορέα που τη λειτουργεί διότι ακριβώς οι διαφορετικές εταιρείες ε, είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει τα χρήματα που θα πληρώνει κανείς για τη χρήση των υποδομών να μπορούν να καταλήξουν στην τσέπη των ανταγωνιστών. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί δεν μπορεί να γίνει καμία, κανένα συμβασμός. Επί της αρχής δεν συμβαζόμαστε στην σύλληψη του συστήματος, απλώς στη διοργάνωσή του μπορούμε να φάνουμε διαλεκτική. Το θέλουμε απλό και διαφανές. Και αυτό που προτείναμε είχε έχει γίνει αποδεκτό και έχει εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο κατά την αναθεώρηση του προηγούμενου πακέτου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την υλοποίηση ακριβώς και να προσέξουμε τι θα κάνουμε με τους φορείς που θέλουν να περάσουν σε ανοιχτό ανταγωνισμό. Θα το συζητήσω όμως ξανά αυτό το ζήτημα. Επίσης για το πεδίο αυτό, για το αυτού του πακέτου, για τις επενδύσεις στις υποδομές και για την διευκόλυνση του, για το μέσο του, της διασύνδεσης της Ευρώπης, του Connecting Europe. Ξέρετε ότι η πρότασή μας ήταν πιο φιλόδοξη. Έχω εργαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών και ξέρω ότι η σχετική μαγειρική είναι από τις πιο περίπλοκες. Όμως, ελπίζουμε ότι για τις υποδομές των μεταφορών θα πετύχει, ελπίζαμε ότι θα περισσότερα. Είναι πολύ μέτρια η αύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις και στην εθνική διανομή των ε, προγραμμάτων, φοβόμαστε ότι θα χαθούν ε, περισσότερα. Ξέρω κύριε Κράμερ και σημειώνω τις παρατηρήσεις σας, τις λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, ανέκαθεν το έκανα αυτό. Θα πρέπει κι εσείς όμως να δεχτείτε ότι υπάρχουν και θετικές κινήσεις. Στα προηγούμενα πανευρωπαϊκά δίκτυα ήδη είχαν γίνει, στα προηγούμενα διευρωπαϊκά δίκτυα ήδη είχαν γίνει κάποιες κινήσεις και τώρα με τις νομοθετικές προτάσεις ελπίζουμε ότι θα εγκριθούν και θα έχουμε μια γερή νομική βάση για να περάσουμε στις μελλοντικέ επενδύσεις. Και να ξεφύγω λίγο από το αυστηρό πλαίσιο της συζήτησή μας εδώ για τις συνδυασμένε μεταφορές. Δεν ε, είναι τα πράγματα τόσο απογοητευτικά όσο λέει ο κύριος Κράμερ. Έχουμε εγκρίνει διάφορες ανακοινώσεις για να προβλέψουμε τις αλλαγές των τιμών στα δίκτυα αυτά. αλλά και εκεί υπάρχει κινητικότητα και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη. Πάντως τα πράγματα δεν είναι τόσο απογοητευτικά. Ιδίω εάν δούμε το πακέτο αυτό καθεαυτό, προβλέπει τη δυνατότητα να υπάρχει ανταγωνισμός μεν, αλλά δικαιότερος, με διαφάνεια και πιο σαφείς κανόνες. Διότι μόνον τότε μπορεί κανείς να έχει ανταγωνισμό δικαιότερο και στον τομέα των μεταφορών. Νομίζω αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα εδώ. Το Αμβούργο και το Βραδεμβούργο δεν είναι ακριβώς η ειδικότητά μου και δεν μπορώ να επηρεάσω εγώ, ειδικά το αεροδρόμιο. Uh, Καλώς ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχω 12 παρακαλώ μιλητές στο κατάλογο μου. Θα σας δώσω ένα τρίλεπτο στο καθένα και μετά 10 λεπτά στον Επίτροπο για να απαντήσει και να κλείσει το θέμα πριν περάσουμε στο επόμενο, την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές. Ζήλε, Ρικέ, Λάιχτφριντ, Σαβισά, Πίρκερ, Μπαχ, Καντσιάν, Φλέκενστάιν, Τρεμόσα, Μπαλσίτης και άλλοι δύο και κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Ζήλε για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Μπράιεν. Συγγνώμη Επίτροπε για την καθυστέρηση. Ε, μερικά σχόλια μόνο να κάνω εγώ προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορα στάδια και σε μια έκθεση ιδιαίτερα που έχει να κάνει με την πιστοποίηση και την έγκριση για την ασφάλεια στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Τώρα, βέβαια δεν έχει μεταφραστεί το κείμενο σε όλες τις γλώσσες, αλλά δεν καλύπτεται η παρούσα κατάσταση. Υπάρχουν και απομονωμένα δίκτυα. Υπάρχουν χώρες όπου η πιστοποίηση δεν κοστίζει τίποτα, αλλά είναι μόνο εθνική και πρέπει να γίνει εντός ενός μηνός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει τέσσερις μήνες κοστίζει, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον θεωρητικά. Υποθέτω και πρακτικά αλλά υπάρχει μια πολύ διάζουσα κατάσταση κάθε φορά και θα πρέπει να φροντίσουμε τελικά όλοι οι ενδιαφερομένοι να καταλήξουν σε ένα καλό συμβιβασμό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για κάποιες ανησυχίες που ακούγονται. Οι εθνικές ενδεχομένως αρχές ασφαλείες ε, υπόκεινται, εντάσσονται στην ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, ΕΡΑ. Άρα αυξάνεται ενδεχομένω ε, το διοικητικό άχθος και η γραφειοκρατία για τις εθνικές αρχές και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, πιστεύω. Πάντως προσβλέπω σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Αν μπορείτε να σχολιάσετε λίγο τις ιδιαίτερες καταστάσεις ε, σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ που τήρησες και το χρόνο. Ο κύριος Ζήκε για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επιτροπό Κάλλας που μας παρουσιάζει αυτή την τέταρτη δέσμη, το τέταρτο πακέτο, το ερώτημα είναι το εξή. Οι Γιατί τα περιβαλλοντικά στοιχεία δεν τα λάβουν, λαμβάνουν επαρκώς υπόψη και δεν αναπτύσσονται όπως θα θέλαμε. Με ένα τόσο περίπλοκο σύστημα σήμανσης και ασφάλειας επίσης. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τάσεις προστατευτισμού και περιορισμού όχι μόνο των φορέων ε, που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές αλλά και των κοινωνικών εταίρων και των εργαζομένων ε, στις μεταφορές και των ε, φορέων ασφάλειας ακόμη κάποιες φορές και των Ευρωπαίων ηθινόντων που προστατεύουν τα εθνικά δίκτυα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Επίτροπε, τρία κεφάλαια, τρεις ομάδες με παρατηρήσεων έχουν να κάνω. Πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό. Ξέρετε ποιε είναι οι προτάσεις του Συμβουλίου στο επίπεδο το δημοσιονομικό για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι ασύμβατες με την υλοποίηση του τετάρτου πακέτου, κυρίως προς τη λειτουργία. Διότι εξηγήστε μας πώς θα μπορέσει ο οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός να έχει νέα ε, οικονομικά μέσα, περισσότερο προσωπικό με έναν ε, μειωμένο προπολογισμό τι θα γίνει με τα μέτρα ασφαλείας, πώς θα υλοποιούνται, θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Έπειτα, η ανάπτυξη των υποδομών, αναφέρθηκαν τα δίκτυα, αλλά και τα διάφορα συστήματα ε, συνδυασμένων μεταφορών και τα ισοδύναμά τους. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα για να δημιουργηθούν. Δεν έχουμε δημοσιονομικά μέσα. Υπάρχει εδώ ένα, μια πρόσκρουση σιδηροδρομική, μια σύγκρουση μεταξύ των προπολογισμού και των σιδηροδρόμων. Έπειτα, δεύτερη παρατηρήση. Εγώ προτιμούσα την προηγούμενη εκδοχή, αλλά με δύο σελίδες εξηγήσεων, ιδιαίτερα περίπλοκες, μιλήσατε για συνδυασμό, αποσυνδυασμό και το καθεξής. Τώρα τα μέτρα που προβλέπονται διασυνοριακά είναι ιδιαίτερα ε, ασαφή και νομίζω ότι το διατακτικό το ίδιο το σύνολο των μέτρων είναι ιδιαίτερο περίπλοκο. Δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη οι επιπτώσει, οι δημοσιονομικέ. Τι γίνεται με την χιονοστιβάδα ποινών που έπεσαν ε, στου περισσότερου από του φόρους των σιδηροδρόμων ήδη από την περασμένη χρονιά. Φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώ οι ροέ οικονομικέ, δεν είναι εκεί το κλεψιά δεν επιτρέπουν την πρόσβαση, δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες προτεραιότητας, ε, ε, κλέβουν και δεν ανταγωνίζονται δίκαια σε άλλα επίπεδα. Τι θα κάνετε για να είναι το σύστημα δίκαιο και να εμποδίσετε αυτού του είδους την κλεψιά που δεν είναι καθόλου οικονομική χρηματική. Και τέλος, Για το θέμα αυτό, εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε μια σαφή και ξεκάθαρη διάκριση, νομίζω ότι θα σας δούμε σύντομα κοντά μας με ένα πέμπτο πακέτο προτάσεων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την απελευθέρωση, ποια η σχέση μεταξύ του πακέτου των σιδηροδρόμων για την απελευθέρωση των κρατικών αγορών και της δημόσιας αγοράς, που είναι κάτι που αυτή τη στιγμή συζητάτε και ποιο το μέλλον του κανονισμού μεταφορών στα πλαίσια και τη εξέλιξη του κανονισμού και τη δημόσια προμήθεια. Επίση, όπω είπαν και πολλοί συνάδελφοι με την κοινωνική διάσταση, τι γίνεται. <clears throat> Θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των 750.000 εργαζομένων στους υδροδρόμου που εξέφρασαν τι ανησυχίε του. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Ολόκληρωσα και θα... Ολοκλήρωσα και θα ξαναεκφραστώ αργότερα. Ευχαριστούμε ο κύριος Λάιχπη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την απελευθέρωση και ε, θα μιλήσω αγγλικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν έγινε κατανοητός ε, όταν μίλησα αγγλικά ε, την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ε, Είπατε ότι οι συντονιστές ε, ασχολήθηκαν ε, σχεδόν ε, με όλα, οπότε εγώ μπορώ να σας ρωτήσω σχετικά με κάποιες λεπτομέρειες. Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τις διάφορες εφαρμογές που υπάρχουν, ξέρω διάφορα συνδρομικά συστήματα όπου ε, ιδιαίτερα κερδοφόρες γραμμές ε, ε, χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν τις λιγότερε κερδοφόρες, αυτές που έχουν λιγότερους επιβάτες. Δεν θέλω να ακούσω ευελιξία από εσά, ότι η Κομισιόν είναι ευέλικτη, θέλω να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις. Σε μια απελευθερωμένη αγορά πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σύστημα. Υπάρχουν αυστηρές εφαρμογές για τις επιχειρήσεις ε, που ε, ασχολούνται με κερδοφόρες ε, διαδρομές ώστε να πρέπει να έχουν και κάποιες μη κερδοφόρες. Επίσης, όσον αφορά το unbundling, την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση ενδεχομένως, δεν καταλαβαίνω. Στην Ευρώπη έχουμε κάποια συστήματα ε, αποδεσμευμένα τα οποία λειτουργούν πολύ καλά. Έχουμε όμως ε, και άλλα που ε, δεν είναι έτσι. Το ελβετικό λειτουργεί εξαιρετικά. Γιατί να το καταστρέψουμε αφού λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντικό αυτό για σας και μία τελευταία ερώτηση που μάλλον δεν είναι ακριβώς ερώτηση, μάλλον έκκληση είναι. Σας παρακαλώ μην ε, μας προβάλλετε το ευρωτανικό σύστημα ως καλό παράδειγμα. Αυτό που είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν καταστροφή νομίζω και στήχησε στον Ευρετανό φορολογούμενο 5 δισεκατομμύρια ε, ευρώ, οι λίρες. Ε, το να ξαναοργανωθεί το σύστημα αυτό. Το βρετανικό παράδειγμα λοιπόν δεν αποτελεί υπόδειγμα. Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στο συνδρομικό τομέα που είχαμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάβησα. Κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα... ήθελα να πω ότι πιστεύω στους σιδηροδρόμους. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να αντικατασταθούν οι σιδηρόδρομοι από ε, δρόμους ε, στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε στους ιδιωτικούς φορείς, τους επιχειρηματίες ε, που στηρίζονται από το κράτος. Είπατε ότι θα υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό θα επηρεάσει τις δημόσιες συμβάσεις. Θα έχουμε κοινούς κανόνες παρά το γεγονός ότι... Ε, ε, άσχετα από το αν ε, οι φορείς αυτοί είναι δημόσιες ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Ε, και η δεύτερη μου ερώτηση, ίσως να μην συνδέεται με το πακέτο αυτό καθεαυτό, αλλά αν το σκεφτούμε ευρύτερα, θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν έχει σκεφτεί να δώσει κίνητρα, τα λεγόμενα καρότα, στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει τα, τις συνδρομικές γραμμές τους. Ε, μπορούμε να δώσουμε κίνητρο στα κράτη-μέλη ώστε να ολοκληρώσουν ε, ε, τις νέες διαδρομές, διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο συνδρομικό χώρο και εσωτερική ε, αγορά, εάν δεν έχουμε ε, κοινέ γραμμές που να μας συνδέουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ μαζί σας σε πολλά πράγματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρόμων, ε, την αγορά που θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Όταν μιλάτε για ασφάλεια και αξιοπιστία, όταν μιλάτε για ένα ενιαίο σύστημα, για δίκαιη πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στις υποδομές, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς ε, το εξής. Ε, στις, ε, στην πρώτη σας παρουσίαση είπατε ότι οι δομές holding μπορούν να διατηρηθούν Στα μέρη όπου κατά την ε, θέση σε ισχύ της πρώτης οδηγίας ε, ήδη υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει αλλαγή εκεί. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα που ήδη λειτουργούν και λειτουργούν καλά δεν ε, θα τα αγγίξετε. Αλλά η αποδέσμευση είναι το non plus ultra για σας, ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ε, για το πακέτο των σιδηροδρόμων. Σας παρακαλώ να μου το εξηγήσετε αυτό, να μου το διευκρινίσετε και ε, Δεύτερον, κατά τις διαπραγματεύσεις του πακέτου για τα αεροδρόμια είχαμε ακριβώς ένα πακέτο και στηρίξαμε αρκετά σημεία, αλλά κάποια άλλα σημεία ε, μας βρίσκουν ε, ε, επιφυλακτικούς, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να αποτύχει όλο το πακέτο εάν το 90% των θεμάτων βρίσκουν κοινή υποστήριξη και το 10% όχι. Μήπως θα ήταν καλύτερο στους συνδρόμους να μην διαπραγματευτούμε το σύνολο του πακέτου, αλλά να εξετάσουμε τα επιμέρους σημεία ε, ώστε να λάβουμε γρήγορη απόφαση όσον αφορά τα σημεία όπου υπάρχει συμφωνία αλλά να μην εξαρτηθεί το σύνολο του πακέτου από το εάν ε, το κάθε μικρό σημείο ε, βρει την υποστήριξη όλων. Νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος της ελεύθερης αγοράς να μην δούμε τη λύση αυτή ως πακέτο, αλλά όπου υπάρχουν καλές λύσεις να πραγματοποιηθούν, ενώ όπου δεν υπάρχει συμφωνία, να προσπαθήσουμε πιο μετά να τα λύσουμε. Κύριε Σμπαχ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι θα έχουμε ασφαλώς ε, επανειλημμένα την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Έχω μια ερώτηση ουσιαστικά που συνεχίζει από τα όσα μόλις είπε ο κύριος Πίρκερ. Αυτή η δέσμη μέτρων για το σιδηρόδρομο εκτελείται ήδη. Ε, ουσιαστικά όλοι ομόφωνα είπαμε ότι προς όφελος της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας, ε, των πελατών, των χρηστών, Θέλουμε αυτά τα θέματα, τα τεχνικά και τη συμβατότητα και τη τεχνική εναρμόνιση να τα προωθήσουμε οπωσδήποτε. Γιατί κατά την άποψή μου εκεί χωλαίνει βασικά ο σιδηρόδρομος. Αλλά τα άλλα θέματα είναι αρκετά επίμαχα. Επανειλημμένα σας έχουμε πιστήσει την προσοχή και διάβασα μια γερμανική ημερήσια εφημερίδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβάλλει αναγκαστικά τον ανταγωνισμό. Μα πώς μπορείτε να το θέλετε αυτό. Είναι πολύ σαφής η θέση του Κοινοβουλίου. Ε, το έχουμε πει εδώ και μήνες. Υπάρχει μια βάση της οποίας μπορούμε να εργαστούμε. Έχουμε αγωνιστεί για έναν ευρωπαϊκό αλλά και εθνικούς ρυθμιστές. Έχουμε αγωνιστεί για τη δυνατότητα ε, ενισχύσεων και χρηματοδότησης και ε, οριζόντιες εγκάρσιες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να τα είχαμε προωθήσει, όπως ε, έχει εξαγγείλει και η Ιρλανδική Προεδρία. Θέλει να προωθήσει τα τεχνικά ζητήματα και είναι καλός αυτός ο τρόπος λειτουργίας και κατά τα άλλα τα υπόλοιπα σε 5 ή σε 10 χρόνια θα μπορούσαμε να τα λύσουμε διαφορετικά έχοντας και εμπειρία. Και όχι τώρα με το ζόρι, μα όλοι οι γνωστοί φορείς είναι αντίθετοι. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ε, δεν συμφωνεί απολύτως. Διαφωνεί το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, έτσι και εδώ τα συνδικάτα, οι εταιρείε οι πάντες. Γιατί αυτή η σύγκρουση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του σιδηροδρόμου. Επόμενη ερώτηση. Μέχρι πριν από λίγους μήνες ε, μιλούσαμε για ένα ανοιχτό μοντέλο, δηλαδή να μην είναι ενιαίο για όλη την Ευρώπη και ομοιόμεθο. Γιατί χάθηκε αυτή η ιδέα, πού πήγε. Γιατί μας είπατε και στην εισαγωγή σας ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις, αλλά και πάρα πολύ διαφορετικά δεδομένα. Ε, ε, κυριαρχικά δικαιώματα, πολιτιστικά, μέγεθος του κράτους, ε, διαδρομή, γραμμή, ε, ακόμα και ιδιαιτερότητες του εδάφους. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα ενός ενιαίου μοντέλου για την Ευρώπη. Εκτός πια αν είναι στενός κορσές. Έχω και άλλες ερωτήσεις και για το προσωπικό, τους εργαζομένους η πρόταση αυτή χωλαίνει, είναι λίγο με βαριά καρδιά. Ε, προτείνεται ε, τι θα γίνει με το τροχαίο υλικό σε περίπτωση εξαγοράς ή τι θα γίνει για την έγκριση των διαφόρων τύπων υλικού, αλλά και το προσωπικό. Όχι πολλά. Πρέπει να σταματήσω εδώ. Ο κύριος Καντσιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω και εγώ ότι Καλό θα ήταν να παραδεχτούμε ότι είναι τεράστιο το έργο σας εδώ, είναι τιτάνια προσπάθεια και για σας λοιπόν και τους συνεργάτες σας συγχαρητήρια όμως θα ήθελα εδώ να αφήσουμε λιγάκι την υποκρισία που και μεταξύ μας καμιά φορά επικρατεί. Λέμε, αν έλεγα μάλλον θέλουμε να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά στην Ευρώπη, νομίζω θα συμφωνούσαμε όλοι από αυτού του στόχου. Όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα, να κοιτάξουμε τι πόρους έχουμε και να καταλάβουμε και πόσο χρόνο διαθέτουμε ε, στη διάθεσή μας και στο σύντομο χρονικό διάστημα. Για όλα αυτά νομίζω τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές ε, ότι θα μας μα πιστεύουν σε αυτού του στόχου μα. Όμω, εάν δούμε πώ εξελίσσονται τα πράγματα, βρισκόμαστε στο τέταρτο πακέτο και αν θυμηθώ τι είχε γίνει με την προηγούμενη συζήτηση για την αναδιατύπωση, εδώ με τις ε, διάφορες ε, εσωτερικές καθυστερήσεις στην Επιτροπή, αυτά που μας είπε ο Επίτροπος για τα τέσσερα είναι ένα πακέτα και ούτω καθεξής, την ολιγορία του Συμβουλίου. Έχω την εντύπωση ότι η υλοποίηση αυτού που θέλουμε και αυτού που πιστεύουμε θα είναι δυσχερέστατη. Δυσχερέστατη και μιλάμε για αρχές, αξίες και όρους που τους ανταλλάσσουμε μεταξύ μας καθημερινά σε διαλόγους σαν να είναι κάτι το δεδομένο. Όλοι εδώ είμαστε υπέρ της διαφάνειας, της αγωνιστικότητας, των πόρων και του σύντομου χρονικού ε, τη σύντομη χρονική υλοποίηση. Όμω υπάρχει δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και στην ε, πραγματική του υλοποίηση. Ω προ του πόρου, ξέρουμε όλοι ποιε είναι οι περικοπέ στον προπολογισμό. Νομίζω ότι πέραν τη προτεραιότητα και των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να εντοπίσουμε, θα χρειαστεί και βούληση. Βούληση για να πάμε προ την κατεύθυνση του ΕΛΚ και των εναλλακτικών πληρωμών σε σχέση με τα τέλη. Mr. Fleckenstein, three minutes, please. Φλέκενστάιν για τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, ήδη αναφέρθηκαν πολλά σημεία για τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και με τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε το στόχο μας. Θα ήθελα όμως να σας θέσω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα της αποδέσμευσης. Ο κύριος Σουγκρός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Στην πρόταση υπάρχει η δυνατότητα υπό κάποιες προϋποθέσεις να διατηρηθεί μια δομή holding. Ε, θεσπίζετε τις προϋποθέσεις. Εσείς ο Δ. Ρίτκε έχει την παραμικρή ιδέα γιατί μία επιχείρηση στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη δομή. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί το, το προβλέπουμε τη δυνατότητα ε, για τη δυνατότητα αυτή. Και τελευταία παρατήρηση, κύριε Πίτροπε, μη μας λέτε ότι δεν υπάρχουν συμβασμοί σας παρακαλώ. Το έχουμε ακούσει αυτό επανειλημμένα και τελικά πάντα βρίσκουμε μια λογική λύση. Σας ευχαριστώ. Thank you, very much, Ο κύριος Μόσα, ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν. Κύριε Επίτροπε, ε, καλώς ήρθατε στο κοινοβούλιο μας. Σε δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Η πρώτη είναι, μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μπορούμε στο τέταρτο πακέτο, στην τέταρτη δεσμή μέτρων, να περιμένουμε ε, κάποιον, να υπάρχει κάποιος Ευρωπαίος ρυθμιστής. Εάν, ε, είναι, εάν ισχύει αυτό, ε, τότε... Νομίζω θα είναι καλό. Πέρσι είχαμε μια συζήτηση για την αναδιατύπωση και ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι συμφωνήσαμε ότι μια ευρωπαϊκή αγορά χρειάζεται και ευρωπαϊκή ρύθμιση και στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, ε, θέμα με το οποίο ασχοληθεί ο κ. Γκρός, ε, ε, αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή και πιέζει για αυτήν. Θέλουμε δηλαδή κάτι παραπάνω από ένα δίκτυο εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Και επίσης όσον αφορά την πρόταση προϋπολογισμού του Συμβουλίου, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για τα βασικά προγράμματα δικτύων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας που στόχο είχε να μα αποσαφηνίσει και τι προθέσει τη Επιτροπή ε, σε σχέση με τι προτάσει για του σιδηροδρόμου ε, και μα αποδείξατε τι έγινε αυτό. Κυρίω όμω θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το καμποτάζ το οδικό. Και είναι τρει οι στόχοι του οποίου συμμεριζόμαστε. Το να υπάρχουν περισσότερε διασυνδομένε μεταφορέ και στο οδικό δίκτυο, να υπάρχει καλύτερη προσφορά και επίση καλύτερη πρόσβαση στι σιδηροδρομικέ υπηρεσίε. Συμφωνούμε σε αυτά. Όμω ε, επιτρέψτε μου κύριε Επιτροπέ να έχω αμφιβολίε για την αναθεώρηση πώς μας την παρουσιάζεται. Ε, φαίνεται να έχουμε μια μαγική συνταγή για να επιτύχουμε και του τρει όχου αυτούς μαζί. Την απελευθέρωση. Και έχω την αίσθηση ότι ξεχνούμε την ουσία και, κάπως βάζουμε το, τα βόδια μπροστά από την άμαξα. Γαλλική έκφραση, ενώ να είμαστε κάπως προδιαστικοί. Δηλαδή έχουμε κάποια δημοσιονομικά μέσα για να επενδύσουμε στις υποδομές σήμερα. Όμως ε, το εφαλτήριο για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα ήταν να επενδύσουμε μαζικά στις υποδομές των σιδηροδρόμων. Όσοι μελέτες και οι αναλύσεις και εθνικές και ευρωπαϊκές δείχνουν ότι έχουμε ανάγκες 300 δις και μετά από τη σύνοδο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου έχουμε ένα προπολογισμό που μειώθηκε κατά 8-9 δις σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής. Ποιες είναι λοιπόν οι πραγματικές μας φιλοδοξίες πέραν της προσέγγισης που εγώ θα την ονόμαζα και δογματική και αδιάλακτη, δηλαδή απελευθέρωση με, τα, με full ταχύτητα. Εδώ ας σκεφτούμε τι συμβαίνει και με την SNCF που έχει έλλειμμα 27 δις τη στιγμή που μιλάμε. Ένα δις λιγότερο το 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε καμία βεβαιότητα όταν κάνουμε την ε, σύγκριση ιδιωτικού ή κρατικού ή τις εθνικές λύσεις που βρέθηκαν. Η, κυρία Επίτροπε, είστε φιλελεύθερος στην προσέγγισή σας. Μπορεί να γίνει και αυτό. Είναι όμως κάπως αυστηρή η προσέγγισή σας. Θέλετε μια συνολική διακυβέρνηση για το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη και επιμένετε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι παντού ενιαίο. Νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ανεξαρτησία του οργανισμού, αλλά όχι δεκαπλασιάζοντας τα κονδύλια, να δούμε τι γίνεται με το κόστος και έπειτα να έχουμε κοινού στόχους, αλλά αφήνοντας και κάποια δυνατότητα ευελιξία στα κράτη-μέλη να έχουμε ε, την ε, διοργάνωση, την οδική και συνδυοδρομική, με διαφάνεια που να μην αδικεί κανένα και με σωστούς οικονομικούς όρους. Επίτροπε, νομίζω ότι αρχίζουμε μια σειρά από συζητήσεις που θα είναι πλούσιες, ελπίζω. Και όπως είπατε και για την διακυβέρνηση, θέλω και εγώ να πω ότι θα ανέκατε πιο διαλλακτικό στη τάση σας, αλλά το ίδιο θα πρέπει να κάνετε και για το θέμα της απελευθέρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο κύριος Βισέπ, ε, στην εισαγωγή σας ε, αναφέρατε ότι ε, στις μεταφορές μειώνεται το μερίδιο του σιδηροδρόμου έναντι των αυτοκινητοδρόμων, των οδικών μεταφορών. Συμφωνώ με τη διαπίστωση, διαφωνώ με το συμπέρασμα που βγάλατε. Μα είναι έλλειψη φιλοδοξίας όσο και πολιτικής βούλησης από την πλευρά των επενδύσεων δηλαδή. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση αυτή. Και ένα σύστημα σιδηροδρομικό ε, που δεν αποδίδει. Εσείς βγάζετε το συμπέρασμα ότι χρειάζεται περισσότερη απελευθέρωση και περισσότερος ανταγωνισμός. Σε καμία περίπτωση μας λέτε ότι οι επιβάτες αναμένουν από το σιδηρόδρομο να έρθει ο ανταγωνισμός. Όχι. Αυτό που περιμένουν οι επιβάτες είναι να φεύγουν και να φτάνουν τα τρένα στην ώρα τους ε, ασφαλή και ανεξάρτητα από τις μετακινήσεις των επιβατών να υπάρχουν τρένα και να μην ε, είναι το εισιτήριο συσχετισμένο με τη διαδρομή, αν η γραμμή δηλαδή αυτή είναι κερδοφόρα ή όχι. Λέτε ότι μετά την έγκριση αυτή τη τέταρτη μέση δεν χρειάζονται πλέον εταιρείε χαρτοφυλακίου. Ε, ε, Υπάρχουν εταιρείε χαρτοφυλακίου που λειτουργούν θαυμάσια, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφάνεια και ανάγκη στη διαφάνεια ε, των ροών των χρηματικών ανάμεσα στην εταιρεία χαρτοφυλακίου και την εταιρεία που διαχειρίζεται ε, την ε, επιχείρηση. Τη λειτουργία δηλαδή των συνδεδρόμων. Και γιατί αυτό να επεκταθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνατότητε που έχει μια εταιρεία χαρτοφυλακή. Σα άκουσα προηγουμένω και δεν αφαιρθήκατε στου εργαζομένου, ε, στου σιδηροδρομικού υπαλλήλου. Επανειλημμένα άκουσα στη συζήτηση που έχουμε σήμερα το απόγευμα ε, το ε, μοντέλο της απελευθέρωσης των εναέριων μεταφορών. Ναι, αλλά αν πρέπει να γίνει με τους ίδιους κοινωνικούς όρους και στο σιδηρόδρομο, οι σιδηροδρομικοί ε, πραγματικά ε, θα πρέπει να φοβούνται το αύριο. Δεν ξέρω τι θα τους ξημερώσει. Αυτά που μας προτείνεται είναι πολύ φιλελεύθερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Ευχαριστούμε κύριε Μπίσσα. Μπορείτε να κλείσετε το μικροφωνό σας. Ο κύριος Ερτούκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άνδρες και οι γυναίκες, κύριε Επίτροπε, έχουν πρόβλημα αυτό τον καιρό. Με την ταχύτητα των διαφόρων απελευθερώσεων δεν μπορούν να το βγάλουν πέρα. Γιατί το λέγω αυτό. Διότι το βλέπω και σε αυτά που μας λέτε. Οπωσδήποτε θέλετε, ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετεί το στόχο, για λόγους ιδεολογικούς θέλετε να απελευθερώσετε με το ζόρι. Γι' αυτό θέλω να σας κάνω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, σε όλη τη συζήτηση και σε όλο το πακέτο το τέταρτο πλέον των σιδηροδρόμων, δεν βλέπουμε πουθενά ούτε παράγραφο, ούτε εδάφιο που να μας δείχνει στη χρηματοδότηση πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα χρηματοδοτούμε τις υποδομές. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι υποδομές να μην είναι από μόνες τους ε, ελληματικές. Πώς σκέφτεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει αυτή τη στραβλή κατάσταση. Γιατί έτσι όπως μας τα περιγράψατε τολμώ να αμφισβητήσω ότι θα το καταφέρουμε. Γιατί, τι συμφέρον θα έχει μια εταιρεία, ας πούμε, μια επιχείρηση, να βάλει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων ως επένδυση στις υποδομές όπως έκανε μέχρι τώρα, αν δεν μπορεί να έχει πλέον ε, έσοδα από αυτό. Γιατί να το κάνει μια εταιρεία, ποιο κίνητρο θα είχε. Θα μπορούσατε να μου το απαντήσετε αυτό παρακαλώ. Ερώτηση δεύτερη. Εάν θυμάμαι καλά, από την πρώτη πρώτου του 2013 έχει τεθεί σε ισχύ αναδιατυπωμένη ε, έκδοση. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπαχ. Προσπαθούμε να επιτύχουμε διάφορα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα πολλά από αυτά ήδη συμπεριλαμβάνονται στην αναδιατύπωση και ισχύουν. Άρα, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε, να δούμε τις συνέπειες, ε, τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα της εφαρμογής και μετά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι στόχος της αναδιατύπωσης ήταν άλλο, δεν το πετύχατε και ε, τίθεστε τώρα να φέρετε για ιδεολογικούς και μόνο μια νέα ρύθμιση. Και αν είναι όλα τόσο ωραία και καλά κύριε Επίτροπε, γιατί αναβάλατε επανειλημμένα τη δημοσίευση της τέταρτης αυτής δέσμης μέτρων ε, για το σιδηρότομο. κύριο κύριος Παλσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα από τη φύση τους, οπότε φυσικό είναι επίσης τέτοιου είδου ε, σχέδια, ε, όπω και αυτά που αφορούν την ενέργεια, να διαλαμβάνουν και πολιτική διάσταση, όχι μόνο οικονομική. Κάθε χώρα πρέπει έναν όγκο εμπορευμάτων να τον ε, διακινήσει μέσω των σιδηροδρόμων. Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό όγκο εισοδήματο εδώ που αφορά όχι μόνο το μετρητό το οποίο συγκεντρώνεται, αλλά και τι θέσει εργασία που δημιουργούνται. Νομίζω λοιπόν ότι σημαντικό εδώ είναι το στοιχείο τη απελευθέρωση. Θα έλεγα, Επίτροπε, στο μέλλον να σκεφτείτε τη μετατροπή των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη. Η από το πρίσμα μιας πολιτικής που να είναι πιο ωφέλιμη και για τους πολίτες. Χάνονται δουλειές εδώ, εταιρείε πτωχεύουν, μετατοπίσεις στι τρίτες χώρες ε, συμβαίνουν συνέχεια. Όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας χάνονται και έχουμε απώλειες των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει όλες οι χώρες να ληφθούν υπόψη ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση, το μήκος ε, του δικτύου, την έκταση του δηλαδή και να σκεφτούμε τι θα γίνει γιατί εδώ έχουμε διαφορετικά τέλη για φορτηγά ή νταλίκες που μεταφέρουν εμπορεύματα στο δικό δίκτυο των χωρών της Βαλτικής Οπότε σα ρωτώ, γιατί εμεί πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Θα χαθούν θέσει εργασία. Λόγω χάρη, 100 θέσει στη δική μα τη χώρα μόνον. Αλλά κάποιοι άλλοι με υψηλά προσόντα, άλλοι τρει σε κάποιο άλλο κράτο μέλο, θα έχουν καλύτερε δουλειέ. Γιατί αυτό να μα ευχαριστεί. Επίση, αν συνεχίσουμε την απελευθέρωση, κάποιε άλλε τρίτε χώρε όπως η Ρωσία, όπου δεν υπάρχουν κανόνες δίκαιου ανταγωνισμού, διαφάνειας και ούτω καθεξής, θα περάσει σε dumping. Ενώ στους δικού μας στους απλώς θα αυξηθούν οι τιμές. Συμφωνώ λοιπόν με την αρχή ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε ώστε, ώστε τα εμπορεύματα να κινούνται περισσότερο μέσω των σιδηροδρόμων από ότι με το δικό δίκτυο, να έχουμε ψηλότερες ταχύτητες για την κίνηση των επιβατών. Σύμφωνοι, για αυτά δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά να σκεφτούμε κάτι άλλο, τις αρχές μας. Αρχές που μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικές αλλαγές και τότε να μας βρείτε περισσότερο σύμφωνος. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σάντερ. Μετά κλείνω τον κατάλογο. Τον είχα κλείσει τον κατάλογο, αλλά θα σας δώσω το λόγο να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την επικία σας. Ε, ζητώ συγγνώμη καθυστέρηση. Έχουμε διάφορα προβλήματα στην Ισπανία. Ε, ζητώ συγγνώμη από τον Αντιπρόεδρο. Ε, θέλουμε ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο να φτιάξουμε, ούτε ε, γερμανικό, ούτε ισπανικό, ούτε γαλλικό. Ένα ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο. Με το διαχωρισμό λοιπόν αυτό την αποσύνδεση του δικτύου από τη λειτουργία. Ε, αυτό αποσκοπήθηκε εσείς. Τώρα είμαστε αισίως στην τέταρτη δέσμη μέτρων με διάφορα στοιχεία, με δύο μεγάλες απουσίες, δύο πράγματα που λείπουν πραγματικά ε, από το πακέτο αυτό. Το ένα είναι η χρηματοδότηση που δεν την έχουμε 8 δις είχαμε, ε, αλλά ήμασταν 12 χώρες λιγότερες προηγουμένως, τώρα έχουμε 13, αλλά είμαστε 27 χώρες συν μία σε λίγο. Ε, μου φαίνεται σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Αλλά ε, δεν υπάρχει και το κοινωνικό υπόβαθρο. Ε, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο εάν δεν αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση στον εξυγχρονισμό και στη διάνοιξη των σιδηροδρόμων ε, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εργαζόμενοι εκεί, άνδρες και γυναίκες. Είναι τελείως ε, ετεροβαρής η πρότασή σας γιατί δεν συμπεριλαμβάνει αυτό το κοινωνικό στοιχείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Επίτροπε. Εντάξει, δεν έχετε και πάρα πολλά εδώ να πείτε. Πολλές από τις απαντήσεις νομίζω ε, ε, μπορεί ε, να καλυφθούν από μία απάντηση. Δηλαδή μία απάντηση σε πολλές ερωτήσεις. Έχετε το λόγο πάντως. Ναι. Πολλές, από τις, πολλές από τις παρατήρησεις έχουν κάνει με την αξιολόγηση των διαφόρων μερών του πακέτου. Και βέβαια Είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε όλε τι συζητήσει, αλλά θα ξεκινήσω από τι τελευταίε παρατηρήσει που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και τι κοινωνικέ πτυχέ. Δεν ε, θέλουμε την απελευθέρωση ε, ω αυτό σκοπό. Το 43% ε, των θέσεων απασχόληση έχουν χάσει συνδρόμοι, στην Ουγγαρία 47%, στην Ρουμανία 60%. Αυτή δεν είναι καλή απάντηση όσον αφορά την απασχόληση. στη μελέτη αντικτύπου υπολογίζουμε ότι 34 ε, εκατομμύρια ε, ε, χιλιόμετρα επιβατών μπορούν να μας φέρουν 14.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η εικόνα. Και πραγματικά έχουμε εκπονήσει πολύ προσεκτικά τις ρήτρες περί κοινωνικού διαλόγου αλλά εάν συνεχίσει παρακμή το σιδηρόδρομο θα χάσουμε και τις θέσεις απασχόλησης και στόχος μας είναι να αυξήσουμε ε, τις ε, υπηρεσίες που παρέχονται στους σιδηρόδρομους. Δεν δέχομαι λοιπόν το επιχείρημα ότι ε, θέλουμε την απελευθέρωση ως αυτό σκοπό. Δεν είναι ιδεολογικό το πακέτο, είναι ρεαλιστικό. Και γιατί αναβλήθηκε το πακέτο αυτό, η δέσμη των μέτρων. Και ένας μήνας είναι τόσο δραματική αναβολή από, τις, από όλη μου την ε, πείρα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το ότι προτάθηκε 19 του και υιοθετήθηκε 30 Ιανουαρίου το πακέτο δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις επενδύσεις, Είπατε ότι η αποδέσμευση είναι κάτι κακό διότι οι ε, επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην ε, υποδομή. Δεν ισχύει αυτό. Ο φορολογούμενος έχει επενδύσει στην υποδομή. Και το 2009 οι επιδοτήσεις ε, μαζί με τις επενδύσεις των φορολογούμενων ήταν 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση αυτή για να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες επενδύσεων. Ε, αυτός είναι επίσης ένας στόχος ε, το, του πακέτου αυτού. Θα υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία στο πακέτο αυτό, γιατί προτείνουμε δέσμη μέτρων ε, γιατί δεν προτείνουμε απλά ε, θέματα διαλειτουργικότητας. Εάν όμως δεν έχουμε ενιαίο χώρο σιδηροδρόμων ή μεταφορών, ε, δεν έχουμε ανάγκη για διαλειτουργικότητα, τότε ο καθένας θα λειτουργεί εντός των συνόρων του και θα μιλάμε για, ευρωπαϊκά, για ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Και εάν θέλετε να έχετε διασυνοριακή διάσταση, και, και πάλι θα πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία δίκαιου ανταγωνισμού Και ακριβώς γι' αυτό δεν δεχόμαστε τα έσοδα από τις υποδομές να στηρίξουν τους ε, οικονομικούς φορείς σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες, για παράδειγμα ε, οικονομικούς φορείς σε άλλες χώρες. Δεν θέλουμε δηλαδή να χρησιμοποιηθούν ε, χρήματα των φορολογούμενων για να δοθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποιον. Και όσον αφορά τους πόρους, Περιμένουμε την, ε, την δική σας απόφαση σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπα, Ο προϋπολογισμός ε, είναι μικρότερος από ό,τι περιμέναμε, αλλά είναι και λιγότερο από, τα, ό,τι χρειάζεται ούτως ή άλλως. Και ε, Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να επενδύσουν στην υποδομή, η εικόνα λοιπόν είναι ευρύτερη. Επίσης, ε, τέθηκε το θέμα σχετικά με την ε, ρυθμιστική αρχή. Προσπαθήσαμε να συνενώσουμε σε ένα δίκτυο τους, ε, τις ρυθμιστικές αρχές, και Υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, βλέπουμε τις λειτουργίες που έχουν οι ρυθμιστές και θα συνεχίσουν να τις έχουν. Ε, όσον αφορά ε, τι ε, μη κερδοφόρε ε, γραμμέ και το κατά πόσο αυτές θα υποστηριχθούν από τα έσοδα από πιο κερδοφόρε γραμμέ, και αν προτείνουμε κάτι. Ναι, πράγματι, προτείνουμε και είναι, έχει να κάνει με την οικονομική ισορροπία. Θέλουμε να βρούμε βέλτιες λύσεις εντό των κρατών μελών και να συνεχίσουμε τι πρακτικέ αυτέ που τα κράτη-μέλη θεωρούν λογικέ. Και δεν ανέφερα πουθενά της, την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύω ότι καλύτερο είναι να βγάζουμε ορθολογιστικά συμπεράσματα και να βλέπουμε τι είναι καλό για τον τομέα των σιδηροδρόμων. Όσον αφορά τα απομονωμένα δίκτυα, ε, το θέμα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά και ε, ο ρόλος ε, των εθνικών αρχών ασφαλείας θα παραμείνει. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δραστηριότητε αυτές. Δεν λέμε τίποτα περί ιδιωτικοποίησης ή μη. Δεν λέμε τίποτα σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορεί να είναι ιδιοκτήτες της υποδομής, ε, Το πακέτο αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση αυτή ούτε τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά θέματα. και δεν ε, θέλουμε να αλλάξει ε, υποχρεωτικά η δομή των εταιριών χαρτοφυλακίου. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά ε, ε τη ροή χρημάτων ανάμεσα στις εταιρείες. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του πακέτου. οι σιδηρόδρομοι βρίσκονται σε άγριο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους μεταφορών. Είναι λοιπόν μεγάλο θέμα ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφορών ε, και είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω αυτό ανα πάσα στιγμή. Αλλά νομίζω καλύτερα είναι να κλείσουμε εδώ όσον αφορά το πακέτο σιδηροδρόμων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε μπροστά μας ενδιαφέρουσες εβδομάδες. Να δούμε. Αποφασίσαμε ποιες ομάδες αναλάβουν ε, τις εκθέσεις για τη δέσμη. Οι ομάδες είναι γνωστές. Ε, προσεχώς θα έχουμε και τα ονόματα των ε, εισηγητών. Για την καθαρή ενέργεια ποιος θα μας το παρουσιάσει εσείς ή ο κύριος Ρούτε. Όχι, είναι τιμωρία ο επίτροπο και θα παραμείνει και για το επόμενο θέμα για την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές. Έχετε και πάλι το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο σημαντικό πακέτο. Εάν φύγετε παρακαλώ αποχωρήστε ησύχω. Όχι εσωτερικέ συζητήσει. Εδώ μία συνεδρίαση μόνο. Εδώ συνεδριάζει η Επιτροπή ε, Μεταφορών και τα πηγαδάκια έξω, παρακαλώ. Λοιπόν, Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη εξαρτάται πολύ από τις εισαγωγέ πετρελαίου για τις μεταφορές και την κινητικότητα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, όχι το χρόνο, την ημέρα δαπανούμε για εισαγωγές ε, και τα μισά πηγαίνουν σε πλοία, αεροπλάνα και ε, γιοταχή και φορτηγά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, προσπαθήσαμε ήδη να κάνουμε την ενέργεια πιο αποδοτική και θα συνεχίσουμε ε, με στόχους φορολόγησης εκπομπών, με έρευνα, ανάπτυξη, αλλά χρειαζόμαστε και μια εναλλακτική στρατηγική αν θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο. 2,5% του ΕΠ μας μας απορροφά κάθε χρόνο ε, εισαγωγή ενέργειας. Λοιπόν, η αγορά αλλάζει γρήγορα και με εναλλακτικέ μορφές ε, μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη ούτε οικονομικά ούτε οικολογικά. Νέες ευκαιρίες λοιπόν και για ε, επιχειρήσεις, για δουλειές και για εργασία των πολιτών. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πακέτο και μια ανακοίνωση που δείχνει ε, μια ολοκληρωμένη στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων ε, με διαφοροποίηση για τις μεταφορές για να ξεφύγουμε από το πετρέλαιο. Ελάχιστη κάλυψη λοιπόν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, και οχήματα που κινούνται με υδρογόνο. Ε, αντίστοιχα ισχύουν και για τα φόρτιγα και ε, για ε, τα πλοία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κύκλος ολόκληρος για ένα πρόγραμμα δράσης και προτείνουμε σταδιακά οι μεταφορές μας να ξεφύγουν από το πετρέλαιο και να περάσουν σε άλλα καύσιμα με μια στρατηγική συνεκτική που προτείνει μια ομαλή μετάβαση σε λύσεις που υπάρχουν σήμερα. Η νομοθετική ε, πτυχή του πακέτου και της δέσμης ε, έχει να κάνει με τη δημιουργία εναλλακτικών δομών ε, που είναι όριμες πλέον να κατασκευαστούν. Και τελικά η αγορά θα αναπτυχθεί με έναν τρόπο συνεκτικό και όχι κατακαιρματισμένο. Η στρατηγική ε, είναι προϊόν συνένεσης και συμφωνιών. Έχουν συμμετάσχει και οι καταναλωτές και ο κλάδος ε, των μεταφορών και των αυτοκινήτων. Ε, υπάρχει μια ελάχιστη κάλυψη υποδομών και πρέπει να περιμένουν έτσι και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για να κανονίσουν την πορεία τους. Τώρα σήμερα η κατάσταση είναι αν έκανε πρώτη η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Το θέμα είναι ότι ε, σήμερα αποθαρρύνονται οι κατασκευαστές να προχωρήσουν τις λύσεις για τις υποδομές υπέρ και των καταναλωτών και των ε, φορέων της αγοράς. Θα κάνουμε οικονομία ε, αν λειτουργήσουμε σε οικονομία κλίμακος. Ε, είναι ένα κλίμα υπέρ των επιχειρήσεων για να μπορέσει και ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει σε μια νέα αγορά. Είναι εδώ πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών για να μπορούν να ανακουφιστούν λίγο τα δημόσια οικονομικά της Ένωσης, να περάσουμε σε, ε, στα κάψιμα του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλά ρυθμιστικά μέσα που έχουν τα κράτη στη τους για να προωθούν τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειάζεται όμως και μία καθοδήγηση από το κράτος να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό σύστημα για να έχουν και νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου ως προς τις προδιαγραφές και το τι ισχύει οι επενδυτές και οι καταναλωτές να έχουν μία ε, σωστή επιλογή με τα λόγου γνώσεως. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ανταγωνισμό με αναδυόμενες χώρες ε, και σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα έχουμε καθυστερήσει. Ολοκληρωνώ λέγοντας ότι με την πρόταση αυτή θα έχουμε ε, και μεγάλη αλλαγή στην νοοτροπία, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κινητικότητα στο μέλλον και το πώς κυκλοφορούμε. Είναι ε, και μια οικονομική αλλά και μια κοινωνική υπόθεση που απασχολεί την κοινωνία δηλαδή και ως προς το οικολογικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εισαγωγή αυτή. Ακούσαμε την προηγούμενη συζήτηση, μάλλον χρειαζόμαστε και εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Γενικά θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω αυτά που προτείνετε. Θα ήθελα να αναφέρω τρία ή τέσσερα σημεία που είναι σημαντικά για μένα. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τις εναλλακτικές πηγές ε, ενέργειας, ιδιαίτερα στις μεταφορές, το θέμα δεν είναι να έχουμε μόνο μία εναλλακτική λύση, να έχουμε διάφορες. Δεύτερον, είναι ωραίο να συζητάμε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και η ανάλογη προσφορά και όσον αφορά την ενέργεια και όσον αφορά την ε, υποδομή. Η, επίσης, τρίτον, η διαλειτουργικότητα είναι και εδώ πολύ σημαντική. Εάν στον τομέα αυτών έχουμε την ίδια κατάσταση με άλλους τομείς, ε, θα διαπιστώσουμε ότι ε, πολλοί πολίτες ε, διστάζουν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για διάφορους λόγους. Πιστεύω ότι ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε άλλους τομείς, όπως ε, για παράδειγμα τις ε, τηλεπικοινωνίες, ε, όπου, τα τηλέφωνα δηλαδή, όπου η Ευρώπη φρόντισε να εισάγει ενιαία πρότυπα, όχι για, μόνο για να πείσουν τους πολίτες, αλλά για να ενισχύσει την Ευρώπη ως τόπο παραγωγής. Και τέλος, με βάση τις εμπειρίες της γειτονικής ε, χώρας ε, στη δική μου, της Γερμανίας, εάν έχουμε κάποια νέα τεχνολογία που ε, ξαφνικά στις εφημερίδες λέει ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους πολίτες, για την υγεία κλπ. Ε, αυτό είναι καταστροφικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι πολίτες να έχουν σωστή πληροφόρηση. Και γενικά επικροτούμε την πρόταση αυτή. Φυσικά θα θέλουμε κάποιες ε, διευκρινήσεις. Νομίζω όμως ότι είναι ο σωστός δρόμος για το μέλλον. Ε, ευχαριστώ κύριε Σαλχαντράου, ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε για την εισαγωγή και την παρουσίαση και την πρόταση. Στην παρούσα φάση θα περιστώ σε γενικές παρατηρήσεις. Και βεβαίω, θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονό ότι επιτέλους έχουμε μια στρατηγική επιχάρτου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη μετάβαση προς ένα στόλο οχημάτων ε, πιο αηφόρο και βιώσιμο. Αλλά χρειάζεται συντονισμό, υποστήριξη από ε, την πολιτεία και η Ευρώπη εδώ πέρα είναι υπαριθμόν ένα ε, πρωταγωνιστής. Ε, μια αγορά καταναλωτών θέλουμε να προκύψει, δηλαδή να γνωρίζουν οι καταναλωτές όλες τις εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις, τις πιο ευφόρες και βιώσιμες και τα μέσα μεταφοράς αλλά και τα καύσιμα. Ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο ε, γνωρίζετε ότι κοστίζει διπλάσια από όσο ένα κανονικό αυτοκίνητο. Ε, δεν μπορούν ε, να ενδιαφέρονται γι' αυτό αρκετοί καταναλωτές όπως έχει σήμερα η κατάσταση. Δεύτερον, σήμερα δεν υπάρχει υποδομή λέμε για να τα ενθαρρύνει όλα αυτά και να μπορούν οι πολίτες να μεταβούν σε πιο αηφόρες επιλογές. Γι' αυτό χρειάζεται να θέσουμε κάποιους στόχους με τεχνική εναρμόνιση και να ξεκαθαρίσουμε διάφορα πράγματα. Η πρότασή σας είναι ε, ουδέτερη τεχνολογικά και καλή καταρχήν. Θα τη μελετήσω, επιφυλάσσομαι. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα συστήματα που προσφέρονται καλύτερα, γιατί δεν έχουν όλα τα συστήματα ε, το ίδιο αποτέλεσμα και τις ίδιες εκπομπές, πούμε, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνεπώς, Ε, πιστεύω ότι χρειάζεται μεν μελέτη, αλλά από πλευρά τη ομάδα μα θεωρούμε ότι βαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Είναι λιγότερο επίμαχη, θα έλεγα, ε, από το προηγούμενο θέμα, το σιδηροδρομικό. Αυτό θα προχωρήσει με περισσότερη συνένεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίαση της πρότασής σας. Τη θεωρώ πολύ καλή και επιγόντως απαραίτητη. Έτσι κι αλλιώς χωρίς υποδομές οι εναλλακτικέ μορφές ενέργειας στις μεταφορές δύσκολα μπορούν να επιβληθούν. Ήδη από σήμερα τι ισχύει. Η, ηλεκτρονική, ηλεκτρική μάλλον κινητικότητα, η mobility, ε, παίζει λιγότερο ρόλο και λιγότερη σημασία από ό,τι στο παρελθόν. Στη Γερμανία Μπορεί κανείς ήδη να κυκλοφορεί και να φορτίζει το αυτοκίνητό του από ένα σημείο στο άλλο, να κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα, αλλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί και τις υποδομές. Και παραμένουν οι καταναλωτές και οι, μάλλον, συγγνώμη, οι κατασκευαστέ και οι αντιπροσωπείες με τα αυτοκίνητα απόλυτα, γιατί ο κόσμο δεν γνωρίζει πώς ε, θα χρησιμοποιεί το δίκτυο. Είναι και το LNG, το υγραέριο, ε, αλλά δεν είναι η μόνη πανάκια η καθαγεσμένη λύση. Αλλά το υγροποιημένο αέριο είναι πολύ ε, καλή, εναλλακτική και όσο και καθαρή μορφή ε, καυσίμου για τα πλοία. Στο Ρότερνταμ υπάρχει αυτή η υποδομή νομίζω, αλλά και στο Ζεμπρούχα αν δεν απατώμε στο Βέλγιο. Και γιατί όχι και για τα φορτηγά, όχι μόνο για τα πλοία. Θα μπορούσε να είναι μια μορφή ενέργειας ε, με αντίστοιχη ε, υποδομή και μετατροπή να ισχύει και για πολλά μέσα μεταφορών. Ε, ρωτώ βέβαια ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Μιλήσατε για ιδιώτες επενδυτές. Μακάρι να τους είχαμε κάθε φορά που τους θέλουμε. Τώρα μιλήσαμε για τη διασύνδεση της Ευρώπης, την περίφημη αυτή διευκόλυνση, μα εκεί τους χάνουμε τους επενδυτές. Πού θα βρούμε επενδυτές για να επενδύσουν αυτή την προσπάθεια. Και ένα τελευταίο, το είπε και ο Ματιογκρός και έχει απολύτως δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα και σωστή πληροφόρηση με το ε10 εγώ Ξέρω και βάζω το κάψιμο ε10 στο αυτοκίνητό μου γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά στην αρχή ήμουνα πάρα πολύ επιφυλακτική στην Αντλία όταν πήγαινα στο πρατήριο να πάρω βενζίνη. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι ισχύει και τι μπορούν να πιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Φυσικά είναι σημαντικό να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε σε ιδεολογική παγίδα. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, ξέρουμε ότι θα έχουμε ακόμα λιγότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πού θα επενδύσουμε. Στο παρελθόν είχαμε κάποιε προόδου. Οι μηχανέ των σιδηροδρόμων χρησιμοποιούσαν περισσότερα καύσιμα ε, πριν 30 χρόνια, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε ε, το θέμα ε, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Από το 1881 Συγγνώμη, με, την, με τις ηλεκτρικές μεταφορές είχαμε ε, ήδη πολύ νωρίς τέτοιο τρένο στην Γερμανία. προσπαθούμε να ε, προωθήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά είναι τόσο μικρή η μείωση των εκπομπών ε, που σχεδόν δεν φαίνεται. θα πρέπει να σκεφτούμε το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών στις μεταφορές ε, που προέρχεται από τις οδικές μεταφορές. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Ο υπουργό Μεταφορών μας είναι πάρα πολύ συντηρητικός. Είπε όμως ότι ε, το 90% των διαδρομών στις ε, γερμανικές ε, πόλεις είναι λιγότερο από 6 χιλιόμετρα. Με, ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα μείωση των εκπομπών. Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε το σύνολο του κύκλου ζωής, όχι μόνο τη χρήση, αλλά και την παραγωγή, και τη χρήση και την ανακύκλωση. Και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ χειρότερα αν κοιτάξουμε το σύνολο του κύκλου ζωής ε, από τα κλασικά αυτοκίνητα. Και τελευταίο θέμα, όταν μιλάμε για ενέργεια θα πρέπει να μιλάμε για, για ανανεώσιμη ενέργεια και θα πρέπει να καταφέρουμε να δεσμεύσουμε τις επιχειρήσεις ε, συντηροδρόμων. Ε, μπορέσαμε στη Γερμανία να ε, αυξήσουμε το ποσοστό των αναλογισμών πηγών ενέργειας από 4 σε 25% ε, αλλά στους σιδηροδρόμους δεν βλέπω καθόλου ηλιακές καταστάσεις ηλιακής ενέργειας μπορούν οι σιδηροδρόμοι να χρησιμοποιήσουν, ε, να εκμεταλλευτούν σωστά τις υποδομές τους. Ε, ίσως θα μπορούσαμε με τροπολογία να το διορθώσουμε αυτό. Πάντως ο στόχος είναι σαφής και να στηρίζουμε εμείς οι πράσινοι. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επιτροπέ. Μια πρώτη παρατήρηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναδούμε τον τίτλο της οδηγίας, διότι ο όρος καύσιμα κάπως με δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εναλλακτική ενέργεια θα πρέπει να λέμε μάλλον περισσότερο από καύσιμα. Είναι πολύ περιοριστικό. Εγώ τουλάχιστον αυτό μπορώ να πω ως πρώτη αντίδραση. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Αλλά και πάλι το μέσο του Connecting Europe Facility, της διευκόλυνσης και την διασύνδεση της Ευρώπης, είναι κάτι που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να δούμε κάποιες μορφές συνεργασίας μεταξύ ενέργειας και μεταφορών, ακριβώς για να προβλέψουμε τις κατάλληλες μεταφορές. Ο ιδιωτικός τομέας επενδύει σε υποδομές που ακόμα όμως δεν είναι αντικείμενο εμπειρίας και οι αγορές δεν μπορεί να χρηματοδοτούν ε, οχήματα τα οποία δεν ε, αξιοποιούνται σε υποδομές που να λειτουργούν. Δημόσια κονδύλια λοιπόν που χάθηκαν ε, με την πρόταση του Συμβουλίου όμως. Αυτά χρειαζόμαστε. Δύο ερωτήσεις λοιπόν κύριε Επίτροπε, Αντιπρόεδρε. Υπάρχουν ε, πολλές πηγές καυσίμων, εναλλακτικής δηλαδή ενέργειας. Μιλήσαμε για το αέριο από βιομάζα. Υπάρχει λοιπόν σε πρώτη φάση το αέριο και τα βιολογικά καύσιμα που μπορεί να προέρχονται από τη γεωργία. Είναι αυτό ένα στοιχείο που δεν μπορούσαμε να καταματρήσουμε, αλλά και κάποια άλλα που προέρχονται από φύκια λόγω χάρη, τα φύκια της θάλασσας. Ε, την ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την ενέργεια, αλλά από την άλλη ότι οι υποδομές που θα χρειαστούν θα είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή γενικόλογη πρόταση όπου στη συνέχεια να δούμε τις νέες μορφές ενέργειας, το να βρεθούν ε, χρήσιμες προτάσεις δεν είναι απλό. Και αυτό σχετίζεται με ένα άλλο ενεργειακό πρόβλημα, της αποθήκευσης της ενέργειας. Αυτό αφορά και την κυκλοφορία και τις ε, μεταφορές και αφορά το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Λόγω χάρη στη Γερμανία γίνεται σημαντική δουλειά και για το υδρογόνο και για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ω πηγή καυσίμων για την ενέργεια, αλλά και για σκοπού ενεργειακή αποθήκευση. Είναι αυτό ενδιαφέρον. Ποια είναι η άποψή σα σχετικά. Διότι θα πρέπει κάπω αυτά τα δύο να τα συνδυάσουμε. Αποθηκεύουμε από τη μια για την ενέργεια, ψάχνουμε ενέργεια για τι μεταφορέ. Πώ θα συνδυαστούν και πώ ε, θα μπορούσαν να τα δούμε από κοινού. Έπειτα για τον εντοπισμό των ε, πηγών που ήδη υπάρχουν. Ε, το αναφέραμε αυτό. Σε κάποιε χώρε υφίστανται κάποιε πηγέ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάποια πρόταση για τον γεωγραφικό εντοπισμό των πηγών των καυσίμων. Ακόμη και αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, ο γεωγραφικός εντοπισμός θα μας βοηθούσε πολύ. Και έπειτα, σε όλη την ε, αλλαγή αυτή που βλέπουμε, την μετακίνηση της, ε, του συνδυασμού των ε, καυσίμων, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης και οι εκπομπές είναι κάτι που μας, θα μας απασχολήσει και συνδυάζεται με όλες αυτές τις προτάσεις θεωρείτε τώρα ότι αυτή η οδηγία είναι μια πρώτη γενική οδηγία, ότι θα πρέπει ήδη να περάσουμε σε απλέ λειτουργικέ προτάσει που να μπορούν να εφαρμοστούν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ απολύτως με τη γενική φιλοδοξία, που είναι και δική μας, να περάσουμε από μια μετάβαση, να περάσουμε σε μια μετάβαση για την ενέργεια στα στι μεταφορέ, αλλά έχω και μια ερώτηση τεχνικού χαρακτήρα από το άρθρο 4 τη οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχουν περισσότερα σημεία επαναφορτισμού με ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ αναφέρονται τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η ανάπτυξή του, αλλά θέλει και να ενοποιηθούν οι τεχνικέ προδιαγραφέ και ε, να υπάρχουν παρόμοιε ε, για όλη την ε, Ευρώπη. Εδώ τι είδους ακριβώς σκέφτεστε γιατί να γίνει αυτή η επιλογή. Ο τύπος α3 ε, αναπτύσσεται, ιδίως στη Γαλλία. Νομίζω κάποιες χώρες είναι πιο προηγμένες ούτως ή άλλως, ε, ως προς τα σημεία αυτά επαναφορτισμού. Το 2015 πιστεύουμε ότι θα έχουμε 5.000 σημεία επαναφορτισης στη Γαλλία. Η επιλογή λοιπόν αυτή, η τεχνική επιλογή, με βάση ποια κριτήρια έγινε. Ευχαριστούμε κυρία Ρόιλ. Κυρία Γιάλα, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ με ενδιαφέρον και ικανοποίηση υποδέχομαι την πρόταση αυτή. Ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Ε, ιδιαίτερα γιατί ε, ακούμε διάφορα νέα κοιτάσματα πετρελαίων και ε, ε άλλα Ε, Μέχρι να μάθω τι έγινε με τα ισπανικά ταξί που έχουν αλλάξει, έχουν περάσει όλο και περισσότερο σε υβριδικά αυτοκίνητα και οι ισπανοί ταξιτζίδες γνωρίζουν αν τους βολεύει ή όχι αυτό το μοντέλο πραγματικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως καλή πρακτική και μια επιτυχία να προβληθεί. Και μέχρι 6.000 ευρώ οικονομία το χρόνο κάνουν γιατί έχουν αλλάξει αυτοκίνητο. Συνήθως είχαν ε, σκόντα και τώρα έχουν το Ιότα υβριδικό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είναι το Ιότα το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε ακόμα αρκετά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ε, και υπάρχει και μεγάλη λίστα αναμονής ε, για τους ευρωπαίους κατασκευαστές. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά τα αυτοκίνητα, κρίμα που είναι το Ιότα Ένα από τα μεγάλα προβλήματα ποιο είναι, οι υποδομές χρόνια ολόκληρα τα λέμε και εγώ ε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω όχι μόνο για τις μεταφορές αλλά και για την ενέργεια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, κινητοποιηθούμε. Εδώ είναι η Γενική Διεύθυνση MOVE, οι μεταφορές. Μα πρόκειται για δίκτυα ε, ενεργειακής τροφοδοσίας και να το πληρώσουν αυτοί που θα βγάλουν λεφτά από αυτή την υπόθεση, που είναι μεγάλες εταιρείες ενέργειας και όχι μεταφορών. Θα πρέπει λίγο περισσότερο να ε, δείξουμε δυναμισμό και να τους υποχρεώσουμε. Ε, τουλάχιστον να κάνουν ε, επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Και τι σχέση έχει αυτό με τις μεταφόρες. Λοιπόν, προσπαθήσαμε ακριβώς να δούμε τι γίνεται με τη συγχρηματοδότηση αυτών των σημείων, των υποδομών, και που θα γίνεται φόρτιση των αυτοκινήτων αυτών. Τι γίνεται με την ασφάλεια όμως, τι γίνεται με τη συντήρηση των νέων οχημάτων. Δηλαδή, ε, δεν θα πρέπει να εκπαιδευτούν νέοι μηχανικοί. Μου το λένε οι οδηγοί ταξί στην Ισπανία, ότι όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που δεν κινείται με βενζίνη ή με δίζελ, δεν ξέρει το συνεργείο να το φτιάξει. Ε, χρειάζεται λοιπόν ε, εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών των συντηρητών. Μπορείτε να μας δώσετε ε, στοιχεία συνολικά ανταλλαγής και πώς θα δοθούν κίνητρα ε, οι κυβερνήσεις ε, που καλούν τώρα σε εξυγχρονισμό των στόλων, των αυτοκινήτων με βοήθειες, ενισχύσεις, απόσυρση, ξέρω εγώ, εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο την απόσυρση και την ανταλλαγή των οχημάτων που να κινούνται με νέα ενέργεια που να μην ρηπαίνει. Εξαρτήσεις, ενημέρωση, προώθηση νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον γιατί έχουν αποτελματωθεί και επενδύσεις όσο και καλές ειδήσει δυστυχώ. Ευχαριστώ ο επιτρόπο. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σα. Η πρότασή μας όντω έχει κάποιες προτάσεις για την ανάγκη παροχής ε, των δεουσών πληροφοριών όμως τέθηκε και το θέμα της χρηματοδότησης και προφανώς δεν το σχολίασα διότι η πρόταση περί χρηματοδότησης βασίζεται σε υπολογισμούς. Θεωρούμε ότι το δίκτυο όπως χρειάζεται θα ε, χρηματοδοτηθεί και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα με 10,5 δις προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποδομές. Αυτό απεικονίζει πόσα μπορούμε να χάσουμε με τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. 40 δις τη χρονιά, 60 κάποιες φορές εξέφνης. Ε, ήταν λοιπόν απλώς μια παρουσίαση αυτής της ε, κατάστασης. Για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη σχετική ιδέα, ναι, είναι μια παλιά ιδέα. Και σαφώς μας ενδιαφέρει να δούμε τον κύκλο ζωής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των σχετικών πόρων. Αυτό έχει να κάνει και με την ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σάντερ, το κατά πόσον συνεργαζόμαστε με την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα. Συνεργασία υπάρχει βεβαίως, συνεισφέρει και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και κυρίως εκείνοι ασχολούνται με τη συντήρηση του νέου, των νέων κατηγοριών οχημάτων. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων από την άλλη αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, αλλά είναι ένα κοινό πρόγραμμα στο οποίο σαφώς θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Ε, και στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων για τα θέματα ασφάλεια. Όσο για τι πηγέ των καυσίμων και όπω είπε και ο κύριο Ρικέτη, θα γίνει με το γεωγραφικό του συντοπισμό. Βεβαίω, η ενεργειακή στρατηγική για την ε, καθαρή ενέργεια για τι μεταφορέ σκοπό έχει να χρησιμοποιεί ευρωπαϊκού πόρου, ευρωπαϊκέ πηγέ ενέργεια, παραγωγού στην Ευρώπη ω εναλλακτική και βεβαίω για να περιορίσουμε και την εξάρτησή μα από το πετρέλαιο. Είναι άκρο σημαντικό αυτό. Αλλά και πάλι, είπε ο κύριος Ρικέ ότι θα πρέπει να κάνουμε σαφέστερες επιλογές για την ενέργεια και τα εναλλακτικέ πηγές. Και είπε η κυρία Μάισερ ότι μία και μόνον λύση δεν μπορεί να υπάρξει, ότι θα είναι δύσκολο να γίνουν σωστές επιλογές των πιθανών πηγών εναλλακτικών ενεργειών. Να αφήσουμε τις αγορές και τα κράτη-μέλη να το καθορίσουν να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και να πάρουν μορφή. Από την Επιτροπή ζητήθηκε πάρα πολύ να πούμε κάτι και για τις προδιαγραφές και για τις υποδομές. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να παράγουν οχήματα, ε, αλλά δεν υπάρχουν χώροι για την επαναφόρτιση, σταθμοί επαναφοδιασμού, κανείς δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Και η βασική πρόθεση της οδηγίας αυτής ήταν ακριβώς ετούτη. Να δώσει κάποιες σαφείς κατευθύνσεις για τη δημιουργία υποδομών. Τελευταίο ερώτημα, αλλά θα μπορούσε ο κύριος Ρόιτε να το σχολιάσει με περισσότερες λεπτομέρειες, αφορά τις ε, ηλεκτρικές πρίζες που είπατε. Είναι δύσκολο το ερώτημα, αλλά στην ε, κινητή τηλεπικοινωνία και το σχετικό δίκτυο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάποιες επιλογές. Ε, τάχθηκε υπέρ μιας λύσης. Αυτό ε, εξυπηρέτησε ολόκληρη τη βιομηχανία γιατί έδωσε σαφείς ενδείξεις για το τι να αναπτύξουν. Το ίδιο χρειαζόμαστε και εδώ. Όταν παράγει κανείς ηλεκτρικό ηλεκτροκίνητα οχήματα. Ήδη υπάρχουν κάποια σημεία επαναφορτισμού. Όμω πρέπει απλώ να γίνει μια επιλογή πρίζα, βίσματο. Και η επιλογή ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων, εντατικών συζητήσεων με του ενδιαφερομένου. Ιδίω με του αυτοκινητοβιομηχάνου και του κατασκευαστέ αυτοκινήτων και άλλος. Αλλά μας είπαν ότι καλό είναι να επιλέξουμε μία μορφή πρίζας. Σίγουρα δεν μπορούμε όλες να τις ε, καλύψουμε, μια επιλογή όμως θα πρέπει να γίνει. Και αυτό για τις απαιτήσει που θα έχουν πια υποδομές για τα κρατημέλη. Ματίας, αν θες κάτι να προσθέσεις, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα, αγαπητοί βουλευτές, κύριε Επίτροπε, νομίζω είπατε σχεδόν τα πάντα στην πραγματικότητα σε κάποια φάση πρέπει κάποιος να επιλέξει ένα πρότυπο, μια προδιαγραφή. Μιλώντας με τους παραγωγούς ε, αυτοκινήτων, ε, μας είπαν ότι το καλύτερο είναι να έχουμε μία πρίζα τα περισσότερα από τα κάτι μέλη. Αυτό προκρίνουν. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ε, ως προς τον αριθμό των κρατών μελών και θα πρέπει να διοργανωθεί μια μεταβατική περίοδος, αλλά δεν στέκει δεν στέκει να υπάρχει μια νησίδα μία πρίζα στην Ευρώπη, ακόμη και για του κατασκευαστέ αυτών των 100 μελών, και να μην μπορούν να εξάγουν στην υπόλοιπη Ένωση εκείνη. Γιατί οι πρίζε είναι διαφορετικέ λόγω χάρη. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τι ΗΠΑ για το είδο πρίζα που θα έχουμε στο όχημα, μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά για την ώρα δεν έχουμε συμφωνήσει για την πρίζα, το βίσμα που θα χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη από την άλλη πλευρά, εκτό. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, πρόταση είναι, θα πρέπει να διοργανώσουμε μια μεταβατική περίοδο, αλλά σε αυτή τη φάση μόνο αυτά μπορώ να πω. Ευχαριστούμε. Νομίζω να πάτε, ότι θα πάτε πιο γρήγορα σε σχέση με το τι είδου φανάρια θα έχουν τα αυτοκίνητα τα τρένα, λόγου χάρη. Σας ευχαριστώ πάντως. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ και τον κύριο Ρόιτε που ήρθατε σήμερα το απόγευμα που μας παρουσιάσατε τη δέσμη για τους σιδηροδρόμους και για την ενέργεια και τις μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επισήμως να διακόψω τη συνεδρίαση. Λύση. Λίγη. επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα στις 18 ε, Μαρτίου στις 3. Στις 3 το απόγευμα. Κλείνει η συνεδρίαση και ευχαριστώ τους ε, διερμηνήσεις.